Αγαπητοί συνάδελφοι, euh, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε αμελητή. δεύτερη Σύνοδος Ολομέλειας ε, της Επιτροπής των Περιφερειών. Καταρχάς, θα σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη με τις εξής αλλαγές. Προτείναμε η γνωμοδότηση του κυρίου Γιάντλα να περάσει από την πρώτη μέρα στη δεύτερη όπως και εκείνη του κυρίου Γιάνσεν, να προταχθεί λίγο, ε, να συζητηθεί λίγο νωρίτερα αύριο το πρωί. Δεν διαφωνεί κανεί. Ωραία. Έχετε αντιρρήσεις σχετικά με τα πρακτικά της προηγουμένης συνόδου. Όχι, πολύ ωραία, εγκρίνονται και τα πρακτικά. Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, γάρδια ε, μία αντιπροσωπεία των ε, δημάρχων που συμμετείχε στην πρόκληση ψηφιακών δήμων που λάνσαρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει 41 πόλεις, δήμους, για να εκπονήσουν ψηφιακές πολιτικές υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των δημοτών. Καλωσορίσατε. Πολύ καλή ιδέα που είχατε να έρθετε στο Ευρωπαϊκό, μάλλον στην Επιτροπή των Περιφερειών, ε, τώρα που έχουμε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω ενωπιών μας την κυρία Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου. Αγαπητή κυρία Κρέτσου, καλωσορίσατε και πάλι στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, σήμερα αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση για πολλές νομοδοτήσεις μετά τη δική σας παρουσίαση για διάφορους κανονισμούς και διάφορες νομοθεσίες που πρέπει να εγκρίνουμε για την επόμενη περίοδο επόμενη προγραμματική περίοδο ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα θα εγκρίνουμε όλες τις νομοδοτήσεις για την πολιτική συνοχή, καθώς και την γνωμοδότηση για την γεωργική πολιτική που συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τι σημαίνει αυτό. Ότι παρόλο που είναι πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, θα έχουμε εγκαίρως μια θεσμική θέση για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πολιτική της συνοχής. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, είμαστε ακριβώς στην ώρα Πέρα από την πολιτική συνοχής, όλες σχεδόν οι νομοδοτήσεις ε, σχετικές με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα εγκριθούν αυτό το διήμερο, ενώ οι προηγούμενες είχαν ψηφιστεί τον Οκτώβρη. Και υπάρχουν ακόμα ορισμένε ας πούμε, αυτή για τον έρασμο που θα έρθει το Φλεβάρι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ολοκληρώνεται τώρα αυτή η προσπάθεια και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για την αγαστή συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εισηγητών μας που ε, είχαν γύρω σήκωση 20 γνωμοδοτήσεις να εκπονήσουν και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέπεια και ε, συνάφεια. Όπως είχα την ευκαιρία να επενθυμίσω, με την έγκριση αυτών των γνωμοδοτήσεων αρχίζει, δεν τελειώνει η ουσιαστική μας δουλειά, διότι τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε οι θέσεις μας να αντικατοπτρίζονται όσο γίνονται περισσότερο στους τελικούς κανονισμούς. Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι πολλές ε, τροπολογίες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετούν και αναγνωρίζουν τη θέση μας. Άρα οι δικοί μας εισηγητές εκ των προτέρων φρόντισαν όλα αυτά να τα προωθήσουν. Σας συγχαίρω. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της Επιτροπής των Περιφερειών και να αυξήσουμε την επιρροή που έχουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι στη ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, απομένει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει στα κράτη-μέλη είδαμε στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και ε, την έννοια των εταιρικών σχέσεων. Υπάρχουν ε, ε, πειρασμοί και τάσεις οπισθοδρόμησης για την πολιτική συνοχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ακούγονται διάφορες λύσεις πολύ απλουστευτικές και ορισμένοι εξακολουθούν να ε, συγχέουν τις έννοιες της απλούστευσης και της ε, συγκέντρωσης της πολιτικής. Ε, απλούστευση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλα να συγκεντρωθούν ξανά κάπου. Και τέλος, για την εδαφική συνεργασία, ακόμα τα κράτη-μέλη διστάζουν. Ας πούμε για τον διασυνοριακό ευρωπαϊκό μηχανισμό. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωρίζει σποδρές αντιδράσεις στο Συμβούλιο. Για όλα αυτά τα θέματα και αφού ψηφίσουμε τις νομοδοτήσεις, ελπίζω ο καθένας από εσά και η κάθε μία να τις αξιοποιήσετε ε, για να τις διαφημίσετε και στα μέσα ενημέρωσης της χώρας σας, ε, αλλά και στους υπουργούς σας υπέρ μιας ε, φιλόδοξης πολιτικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο, για να μην πω το σημαντικότερο που καλούμαστε να επιτελέσουμε τους επόμενους μήνες. Επίσης, είναι το έργο που χωράει περισσότερη βελτίωση. Υπολογίζω στον καθένα από εσάς, σε κάθε εθνική αντιπροσωπεία, σε κάθε ομάδα, για να μπορέσουμε πραγματικά να ε, διακηρύξουμε τις θέσεις μας. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε και πάλι με τους ηγητές μας και την αρμόδια επίτροπο για τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής. Κυρία Κρέτσου, αγαπητή Κορίνα, έχετε το λόγο για να μας κάνετε μια εισαγωγή πριν τη συζήτηση με τα μέλη μας. Thank you Ευχαριστώ πολύ, Καρλ Χάιντς. Πρόεδρε Καρλ Χάιντς Λάμπρετς, αγαπητοί. Καλησπέρα σας και με μεγάλη μου χαρά. Σήμερα είμαι εδώ κοντά σας. Είναι σημαντική η συμβολή σας όσον αφορά την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον της ε, πολιτικής μας συνοχής, των περιφερειών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια. Ιδίω για την ταχύτητα με την οποία έχετε συντάξει αυτές τις ισορροπημένες ε, εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε τα προγράμματα έτοιμα να τρέξουν θα πρέπει να έχουμε αυτούς οι οποίοι έχουν τον ρόλο των πιλωτικό, τον ρόλο του παραδείγματος προς μίμηση, τους pace και για τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πάλι ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Ιδίως δε να ευχαριστήσω τον συνασπισμό της συνοχής. Μάρκο, Καρλ Χάιντς, σας ευχαριστώ για αυτές τις προσπάθειες που από κοινού έχετε καταβάλει. Γιατί ε, πρόκειται για την πιο δύσκολη φάση αυτής της προετοιμασίας του πολιτού πλήσιου. τη φωνή στις πόλεις και στις περιφέρειες. Μια φωνή που αντιστοιχεί στην πεποίθησή του στην Ευρώπη, μια φωνή βοήθειας για τα όσα και εμείς πρεσβεύουμε για την Ευρώπη. Καμία περιφέρεια δεν θα μείνει ουραγός. Και πάλι ακούγεται η φωνή σας και με τις γνωμοδοτήσεις σας μας βοηθάτε, μας στηρίζετε όπως το είπε και ο Καρλ Χάιντς και πρόκειται για τρεις βασικούς τομείς. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις εταιρικές σχέσεις γιατί η επιτυχία της περιφερειακής πολιτικής βασίζεται στους περιφερειακούς εταίρους, περιφερειακές αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, το πόσο θα πιάσει τόπο η πολιτική επιτόπου. Αυτό χρειάζεται. Θα πρέπει να υπάρχει απλούστευση. Και αυτό το κάνετε εσείς με το ότι ξέρετε τι συμβαίνει επιτόπου και ε, όλα αυτά με το δυναμισμό σας, την αποφασιστικότητά σας να βελτιώσετε τη ζωή του κόσμου στις περιφέρειά σας και πάλι Ευχαριστούμε για αυτή την αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική που μόνο με ισχυρούς εταίρους είναι εφικτή. Επίσης, την εταιρική συμφωνία που καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται να έχουμε μια στρατηγική έποψη των πραγμάτων και συντονισμό μεταξύ ταμείων, προγραμμάτων. Χρειάζεται να συνομιλούμε με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς ε, παράγοντες την κοινωνία των πολιτών. Ε, γι' αυτό και οι εταιρικέ συμφωνίες για όλα τα κρατημέλη χρειάζονται. Είναι κάτι το αναγκαίο. Άσχετα από το πόσα προγράμματα υπάρχουν, άσχετα από το τι πρικοδοτήσεις υπάρχουν, δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωράνε κατά τη γνώμη μας. Και η θέση μου κατά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ακούστηκε ξεκάθαρη. Προτείναμε να υπάρξει κάποια εξαίρεση όσον αφορά την υποχρεωτικότητα των εταιρικών συμφωνιών. Και όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στυλώσει τα πόδια. Δεν μετακινείται από τη θέση της. Χρειαζόμαστε για όλα τα κατημέλια στρατηγική. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κρατημέλη πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Επίσης, συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει τοπική ανάπτυξη ο κόσμος, οι πολίτες, οι τοπικοί, για τις τοπικές ανάγκες. Συνεργασία με αυτούς λοιπόν, για το λαό, με το λαό να γίνονται όλα αυτά. Αυτό δεν είναι μία απλή διακήρυξη, απλά λόγια. Είναι μία πολιτική δέσμευση. Πρόκειται για τον στόχο υπαριθμών πέντε της πολιτικής μας. Και έτσι θέλουμε αυτή η δέσμευση να υλοποιηθεί και έχουμε διάφορα μέσα διάφορα μέσα για την επικράτεια οπότε υπάρχει το, η πρωτοβουλία για τις πόλεις για την ανάπτυξη στην πολιτική συνοχή και υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης τη Υπέθρου και έτσι θέλουμε οι περιφέρειες να χειραφετηθούν, οι πόλεις, ε, ο κόσμος ε, εκεί που μένει για το τι κάνει η Ευρώπη για αυτούς, όλοι να ξέρουν και κάτι άλλο τώρα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το θέμα έχει σχέση με την υποχρεωτικότητα αυτών των συμφωνιών. Ε, το ζήτημα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Έχουμε το 5 συν 2 του προγραμματισμού. Ξέρω ότι διατηρείτε κάποιες επιφυλάξεις, προβληματισμούς έχετε, αλλά θέλω αυτά να τα ακούσω, να μου τα πείτε τώρα, σε λίγο την ώρα που θα έχω την τιμή να ακούσω τις απόψεις σας. Αλλά να σας εξηγήσω πώς βλέπουμε τα πράγματα. Γιατί θέλουμε να υπάρχει αυτό το περιθώριο ελιγμών, αυτή η ευελιξία. Ξέρω ότι επί της αρχής συμφωνούμε. Θέλετε πιο ευέλικτη πολιτική η πολιτική αυτή να καλύπτει τις ανάγκες όπως προκύπτουν, χωρίς να παρεμποδίζονται τα πιο μακρόπνοα σχέδιά μας. Είδαμε τι έγινε στο παρελθόν. Είχαμε την αξιολόγηση της επίδοσης. Αυτό ήταν για δύο προγραμματικές περιόδους, η περίοδος προγραμματισμού τέλος πάντων. Αυτό απέδωσε. Είχαμε και τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση στα πέντε χρόνια. Και την τελευταία τετραετία έμαθα ότι δεν είναι δυνατόν 7 χρόνια πριν κανείς να προβλέψει τι θα προκύψει. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Πάντως, για να κλείσω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την βοήθειά σας σε τόσους τομείς. Τα τελευταία αυτά δύσκολα χρόνια που είχαμε την προετοιμασία του επομένου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Την εταιρική συμφωνία και πάλι σας λέω ότι περιμένω σε απόψεις σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Χωρίς άλλη καθυστέρηση μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να σε υπενθυμίσω ότι αυτή τη φορά πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες φορές θα πρέπει να είμαι πολύ, πάρα πολύ αυστηρός με τον χρόνο αγόρευσης. Διότι δεν θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλα τα σημεία της ημέρης της διάταξης ούτε για σήμερα ούτε για αύριο. Έχουμε 15 εγγεγραμμένου ομιλητέ. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση μέχρι τις 4 και 4. Α είστε λοιπόν αρκετά σύντομοι στι παρεμβάσει σα, αλλά προφανώς θα πρέπει να εκφράσετε την άποψή σας. Ας ε, ξεκινήσουμε με τον Μικαέλ Σνάιντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι σήμερα σημαντικό αυτό το βήμα σταθμός στην κοινή πορεία. Το 2016 αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε για την περίοδο μετά το 2021. Το Μάιο του 2017 γνωμοδοτήσαμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Εδώ σε αυτή την αίθουσα το ψηφίσαμε. Ε, και ε, έτσι δημιουργήθηκε ο συνασπισμός ε, για τη συνοχή. Ήταν κάτι το αυθόρμητο και στέφτηκε με τεράστια επιτυχία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάντα ήμασταν σε στενή συνεργασία και επαφή και με εσάς και με ειδικούς από τη γενική σας διεύθυνση. Και το γεγονός ότι οι δικές σας προτάσεις για τα διορθωτικά ταμεία που δημοσιεύσατε φέτος το Μάη έχουν συμπεριλάβει σε πολλά σημεία δικές μας προτάσεις. Αυτό τι αποδεικνύει, ότι είναι το αποτέλεσμα και καρπός μιας μακροχρόνιας εντατικής και καλής συνεργασίας. Σας ευχαριστώ και είναι προς το συμφέρον και των δύο. Ε, αυτό. Άρα, καταρχήν καλωσορίζουμε τις προτάσεις σας, ιδιαίτερα ε, το γενικό κανονισμό. Βεβαίως, υπάρχουν και κάποια σημεία όπου λέμε ότι χωράνε και βελτίωση. Ε, να σας αναφέρω μερικά σε αυτή τη γενική συζήτηση. Απαντώ στην ερώτησή σα, 5 συν 2, γιατί έχουμε αντιρρήσει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το, συν 2 και, ε, το 5 συν 2 και με την ε, ευελιξία. Απλώ είναι ασαφεί οι προτάσει και οι κανόνε Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε και δεν επιτρέπεται ε, να γίνει είναι μετά από μια πενταετία να ξαναρχίσουμε από το μηδέν για την επόμενη διετία. Τουλάχιστον για τα δύο τελευταία χρόνια θα πρέπει ενδεικτικά να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε τα κονδύλια να απορροφηθούν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ε, και άλλα σημεία μεμονωμένα. Καλά έχετε προβλέψει μια ασφαλιστική δικλίδα, ένα δίχτυ ασφαλείας. 76% ε, κανένας δεν πέφτει πιο κάτω, αλλά το πεδίο αναφορά είναι το εθνικό επίπεδο. Και σε πολλές περιπτώσεις στα κράτη-μέλη αυτό δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι δίκαιο, γιατί οι περιφέρειες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, στη Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και αλλού. Άρα το 76% δίκτυα ασφαλείας ναι, αλλά το επίπεδο αναφοράς να είναι το περιφερειακό, όχι το εθνικό. Όπως ορίζεται σήμερα ε, το περιφερειακό επίπεδο να μην είναι καμία περιφέρεια κάτω του 76%. Στη συνέχεια, συνυπευθυνότητα, συγχρηματοδότηση. Κάνατε πολλέ προτάσει για να μειωθούν οι συντελεστέ συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ ανήκω σε μια παράταξη και μάλλον και σε μια περιφέρεια που έχει και δημοσιονομικές εξουσίες ε, δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Θα πρέπει να τηρήσουμε και αυτό το φρένο που έχουμε για την ανάληψη χρεών. Πρέπει να εξηγιάνουμε τον προπολογισμό μας στην περιφέρεια. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε το συντελεστή τη χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες που είναι σε μετάβαση. Δεν θα πρέπει να πέσει κάτω του 70% η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τρίτον, ε, δεχτήκατε την πρότασή μας να έχουμε και άλλους δείκτες εκτός από το ΑΕΠ και συμφωνούμε. Αλλά υπάρχουν κάποια δημογραφικά προβλήματα. Που, ε, αυτός είναι ένας δείκτης που δεν λαμβάνεται υπόψη αρκετά. Θα πρέπει πολύ περισσότερο να τα σκεφτόμαστε αυτά για τις περιφέρειες. Τα δημογραφικά προβλήματα εμποδίζουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και ακριβώς αυτό είναι στο κέντρο της πολιτικής συνοχής να αποφευθεί. Σας παρακαλώ λοιπόν βάλτε και το δημογραφικό δείκτη ως επιπλέον. Και ένα τελευταίο. Έχετε κάνει καλές προτάσεις για την μείωση της γραφειοκρατίας στη διοίκηση. Αυτά που ακούω από τις διαπραγματεύσεις μου έχουν βάλει ψήλους στα αυτιά. Έχω την εντύπωση ότι ε, το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη ε, ξαναβάζουν στη διαπραγμάτευση αυτό που αφαιρέσατε εσείς. Και έχουμε την ίδια γραφειοκρατία που εμείς οι δυο θέλουμε να αποφύγουμε. Έκκληση απευθύνω στους διαπραγματευτές. Μη φορτώνετε πάρα πολύ τη βάρκα. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Επόμενος ο μιλητής. Κατιούσα Μαρίνη. Ομιλήτρια Κατιούσα Μαρίνη. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Σε ευχαριστώ Κορίνα. Για μία ακόμα φορά μας δείχνεις με την παρουσία σου εδώ σήμερα που στην Ολομέλειά μας θα συζητήσουμε όλες αυτές τις γνωμοδοτήσεις όσον αφορά τον προγραμματισμό των διαρθρωτικών ταμείων. Μας δείχνεις λοιπόν ότι είσαι πάρα πολύ κοντά μας και ότι είσαι πάντα σύμμαχος τελικά των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων μαζί με πάρα πολλούς άλλους σημαντικούς παράγοντες δημιουργήσαμε αυτή τη συμμαχία της συνοχής και είχαμε και εσένα στο πλευρό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική συνοχή αποτελεί το πιο θετικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοντά στους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Απευθύνεται άμεση πολιτική αυτή σε πολίτες, σε επιχειρηματίες, σε ηθήνονται σε τοπικό επίπεδο. Εκπροσωπώντας α, τη σοσιαλιστική ομάδα, πρέπει να αναφέρω κάποια σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την τελική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνούμε με την αρτεκτονική την οποία προτείνατε που καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρείται την αρτεκτονική αυτή σε τρία επίπεδα όσον αφορά την επέμβαση των ταμείων της πολιτικής συνοχής. Έχουμε μία προσέγγιση η οποία, όπως είπες και εσύ, θα πρέπει πραγματικά να λαμβάνει υπόψη της τις συμφωνίες εταιρική σχέσης που υπάρχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βλέπει επίσης η προσέγγιση αυτή πραγματικά ποια είναι η σχέση μεταξύ τοπικού και εθνικού επίπεδου, κεντρικού επίπεδου. Είχαμε θέσει όμως και κάποια σημεία, τα οποία μπορείτε να δείτε και στην τελική γνωμοδότηση την οποία θα πρέπει να εγκρίνουμε, ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο, ανεφέρετο τμήμα του πλαισίου προγραμματισμού για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αν δεν υπάρχει η κοινωνική διάσταση που έχει να κάνει με συγκεκριμένε υπηρεσίε, ιδίω στον τομέα τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να ληφθούν υπόψη όλε οι προσπάθειε που καταβάλαμε τελευταία χρόνια, προκειμένου να μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματικά να φουγκραζόμαστε τι πραγματικέ ανάγκε, όπω αυτέ απορρέουν από του τοπικά και περιφερειακά ευθύνοντε. Λέμε στη γνωμοδότησή μας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμείνουμε σε κάποια σημεία βελτίωσης ε, του συστήματος. Πρώτον, να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερο τους τοπικούς και περιφερειακούς ηθήνοντες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης έχουμε και κάποιες ανησυχίες τις οποίες θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας. Βλέπουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο προγραμματισμού το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξαφνικά βρίσκεται εκτός του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις περιφέρειές μας. Για όλες εκείνες δηλαδή τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες, οι οποίες έχουν πιο αγροτικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά υπαίθρου και νομίζω ότι όσον αφορά το ζήτημα τη διοίκηση και τη γραφειοκρατία, δεν εξαρτώνται όλα από την Ευρώπη. Η διοικητική απλούστευση είναι σαφώ πάρα πολύ σημαντική και προφανώ θα πρέπει αυτή να απορρέει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό εκτιμούμε και τι δικέ σα προτάσει. Θέλουμε προφανώ να απλουστεύσουμε τι γραφειοκρατικέ αυτέ διαδικασίε που προβλέπονται όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να είναι πιο εύκολη πρόσβαση στου πόρου, αλλά και προκειμένου οι πόροι αυτοί να μπορούν να απορροφώνται καλύτερα και πιο γρήγορα. Και τελευταίο μήνυμα, το είπε και ο Πρόεδρος και το επαναλαμβάνω και εγώ, η γνωμοδότηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τελικό προορισμό. Είναι μόνο αφετηρία για μία καλύτερη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα θέλαμε πραγματικά η πολιτική συνοχή να μην αποτελεί μόνο αντικείμενο διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κεντρικών, κυβερνήσεων, αλλά θέλουμε περισσότερο διάλογο και μεγαλύτερη συνεργασία με το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα θέλαμε λοιπόν να εισακουστούμε περισσότερο στο πλαίσιο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, κύριε Επίτροπε Θέλω να σας συγχαρώ για την καλή δουλειά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονώντας αυτές τις προτάσεις. Πάρα πολύ σκληρή δουλειά έγινε και το ξέρω σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνογή και βλέπουμε ότι έχουν γίνει και πολύ μεγάλα βήματα προς την απλούστευση. Αυτό το βλέπετε από την υποστήριξη που έχετε στις προτάσεις σας από τους εταίρους στις περιφέρειες. Είναι πολύ σημαντικό να ισχύει για όλες τις περιφέρειες αυτό. Και για τις επαρχίες της Ολλανδίας που είναι η πατρίδα μου. Και πραγματικά βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εταιρική σχέση και οι συμφωνίες και εσάς. Και βλέπουμε το ρόλο των περιφερειών, των επαρχιών, των πόλεων και είναι ένα από τα θέματα ε, που αναφέρω και στην έκθεσή μου για το Ταμείο ανάπτυξη της Υπέθρου και ε, για το Ταμείο Συνοχής. Ιδιαίτερα οι θεματικές συγκεντρώσεις που θέλουμε ε, να γίνονται σε επίπεδο περιφερειών και να παραμείνουν ισχυρέ οι περιφέρειες. Επίσης θέλουμε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκτέλεση ε, του προγράμματος, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για τη μετανάστευση και την εσωτερική, την ενδοευρωπαϊκή. Γιατί ξέρετε ότι ε, φεύγει ο πληθυσμός από την Ανατολική Ευρώπη ε, και παρατηρείται και κάποια απερίμωση εκεί στις περιφέρειες. Η νομοθεσία είναι σημαντικό να γίνει πολύ ε, απλούστερη και να είναι σε θέση οι υπάλληλοι που καλούνται να την εφαρμόσουν να το κάνουν, να τα γνωρίζουν αυτά τα θέματα. Σε συζητήσεις που είχα σε όλη την Ευρώπη για τη γνωμοδότησή μου βλέπω ότι υπάρχει συναντήληψη για τις περιφέρειες. Είτε είναι ε, το εμπορικό επιμελητήριο, ε, στην Klagenfurt της Αυστρίας που έχει και την Προεδρία, είτε όποια άλλη ε, περιφέρεια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι συμφωνούν. Αλλά βέβαια η πολιτική συνοχή υφίσταται πιέσεις από το ρόλο που παίζουν τα ίδια τα κράτη-μέλη μας εκεί. Εμείς ως Ευρωπαϊκές Περιφέρειες είμαστε στο πλευρό σας μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αγώνα να παραμείνει μια σωστή αξιοπρεπής πολιτική συνοχής και στο μέλλον και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο να σας βοηθήσουμε, το ακούω. Μέχρι τότε, καλή τύχη στον τριμερή διάλογο για αυτό το δύσκολο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Αντουανέτ Μομπερσούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε, Κύριε Επίτροπε, έχουμε να γνωμοδοτήσουμε διάφορε προτάσει σα όσον αφορά για την περίοδο 2020, όσον αφορά την πολιτική συνοχή και η πολιτική μα ομάδα. Σα βεβαιώ ότι εργάστηκε όχι μόνο για να έχουμε κάποιε συνεπεί νομοδοτήσει για μια τέτοια δυναμική, αλλά επίση θέλουμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο είναι αυτό το οποίο θέλει ο κόσμο. και θα πρέπει να πετύχουμε σε αυτό το στόχο το 2020 και θα πρέπει να δούμε από σήμερα, από τώρα, πώς θα πείσουμε όχι μόνο τα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να πείσουμε του ευρωσκεπτικιστέ για το ότι η Ευρώπη είναι και για αυτούς και όχι εναντίον εκείνων. Γιατί επίσης έχουμε ε, αυτό το οποίο έγινε την ε, Δευτέρα στο Κοινοβούλιο ε, σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Αλλά αυτό αφορά επίσης και τις αρχές, τις βάσεις Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις δύο άλλες πτυχές σε σχέση με την δαφική συνεργασία. Αυτό να γίνει για την απότερη περιφέρεια και επίσης να έχουν κάποια σχέδια καινοτομία διαπεριφερειακά. Οπότε αυτό το, το, τετράμινο ε, όλα αυτά έγιναν και χτες καταλήξαμε ότι αυτή την πτυχή Interreg Ευρώπη είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στο πνεύμα της εδαφικής συνεργασίας και έτσι ε, μετραχόμαστε κάποιες ε, συγκεκριμένες ε, εμπειρίες και αυτό αποτελεί επίσης μια προσθεμένη αξία. Όμως οι διαμεθοριακές θαλάσσιες περιοχές έχουν κάποιες επιφυλάξεις γιατί εκεί στο ΝΑΤΣ 3 υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις γειτονιάζουσες θαλάσσιες περιοχές στην ε, διάσκεψη που έγινε αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα κριτήριο συγκέντρωσης του πληθυσμού για μια ζώνη 25 χιλιόμετρων για αυτή την ε, ζώνη ε, κατά ξηράνη και έτσι να εμπλακούν αυτοί οι τοπικοί παράγοντες αμφιβολίες και αβεβαιότητες. Τι λέτε κύριε Επίτροπε, δεν θα πρέπει αυτό να γίνει στην επικράτειά μας, δηλαδή ό,τι δουλεύει να το κρατήσουμε και να αξιοποιήσουμε ό,τι μας ε, ενώνει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα τον λόγο έχει ο Μπουκ Άλντσα. Ευχαριστώ ε, πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Κρέτσου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη δήλωσή σας, κυρίως για την αφοσίωσή σας στην πολιτική συνοχής. Κάθε φορά το βλέπουμε όταν έρχεστε. Εγώ ε, είμαι από τη Μεθόριο ε, Γερμανίας Ολλανδίας και τοπικός άρχοντας και χαίρομαι για τα όσα προτείνεται ε, και για την διασυνοριακή συνεργασία. Διότι στο κάτω-κάτω αυτό αφορά 30% των κατοίκων τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Προσωπικά είμαι συντάκτη νομοδότηση για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ε, τον κανονισμό για ένα μηχανισμό διασυνοριακής συνεργασίας ε, έτσι ώστε να ξεπερνάμε πιο γρήγορα νομικά και διοικητικά εμπόδια και προβλήματα και να τα λύνουμε. Οι περιφέρειες το βλέπουν θετικά αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιφέρειες και πόλεις θα έχουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας και ζητούν αυτό το εργαλείο να υλοποιηθεί. Με την χρηματοδότηση ε, Interreg ε, και τις άλλες πρόνοιες για την διασυνοριακή συνεργασία και την περιφερική ανάπτυξη. Ανησυχούμε, Πρόεδρε, για τη συζήτηση που κάνουν στο Συμβούλιο των Υπουργών, γιατί βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη είναι διστακτικά και απρόθυμα. Σας παρακαλώ φροντίστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει αυτή η υπόθεση με τρόπο επικοδομητικό, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το εργαλείο για να υπάρξει ουσιαστική πολιτική συνοχή και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Εμίλ Μποκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Κρέτσου, Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Επίτροπε για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει προκειμένου να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής σε όλες τις γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμερίζομαι το δικό σας το, άρωμα, το όραμα για μια πολιτική συνοχή για όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κανείς δεν θα μένει πίσω. Ορισμένες ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση ω δήμαρχο τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Ρουμανία, είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με πολλού πολίτε, με πολλού νέου συγκεκριμένα, οι οποίοι μου είπαν ότι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τη χρησιμοποίηση κάποιων ευρωπαϊκών κονδυλίων γιατί η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα γραφειοκρατική, πολύπλοκη, χρονοβόρα. Από την άποψη λοιπόν αυτή, έχοντα υπόψη το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ποιο είναι το μήνυμα που θα στέλνατε εσεί στου νέου αυτού που θέλουν να κάνουν αίτηση για ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά αποθαρρύνονται από τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε. Δεύτερο ερώτημα. Όσον αφορά το N συν 2 ή N συν 3. Εγώ είμαι υπέρ της αρχής 1 3, γιατί θα γνωρίζετε ότι καθώς εμείς μπήκαμε αργότερα στις διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς θέλουμε να απορροφήσουμε όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Αν εξ αρχής λοιπόν μπορούμε να έχουμε και για μας την αρχή νύνση 3, αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην πράξη τα κονδύλια. Τρίτη ερώτηση, μια συμβουλή που θα ήθελα μάλλον από εσά. Έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό εργαλείο την πρωτοβουλία για τις πόλεις, την αστική πρωτοβουλία. Ως δήμαρχος, αλλά και για τους υπόλοιπους συναδέλφους στην Επιτροπή των Περιφερειών, τι μας συμβουλεύετε, πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για να χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά το νέο αυτό εργαλείο, προκειμένου να ασφαλίσουμε κονδύλια από την αρχή, από την πρώτη φάση χρησιμοποίησής του. Και μια παρατήρηση. Αν δεν κάνω λάθος, η πολιτική συνοχής άρχισε να εφαρμόζεται με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1973 ή μάλλον ήταν προσχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά μένει πολιτική συνοχή. Ποια είναι η μαλλον ηταν προσχωρησε του Ηνωμένου βασιλειο στην ευρωπαικη ενωση αποχωρει το ηνωμενο βασιλειο αλλα μενει πολιτικη συνοχη ποια ειναι η δικη Σα άποψη όσον αφορά το μέλλον τη πολιτικη συνοχη σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο τη αποχωρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ιζαμπέλ Μπουλινό έχει τώρα το λόγο. σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, Εξ ονόματος της ομάδας των σοσιαλιστών σας ευχαριστούμε ειλικρινά γιατί πάντα ήσασταν στο πλευρό των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Πραγματικά μπορούσαμε να βασιστούμε στη δική σας την και τη δέσμευση την οποία γενναιόδωρα κάθε φορά μας δίνατε προκειμένου να έχουμε μια πολιτική συνοχή πραγματικά για όλα τα εδάφη, για όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και διέπει η ιδέα αυτή την γνωμοδότηση των Κατιού Χαμαρίνη και του Μικαέλ Σνάιντερ για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλε οι περιφέρειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύονται από μια πολιτική συνοχή, μια επενδυτική πολιτική που να απευθύνεται σε όλε τι περιφέρειε. Τον έχουμε περιορισμού για συγκεκριμένε μόνο περιφέρειε όσον αφορά αυτή την πολιτική ενέχει πάρα πολλού κινδύνου, δημιουργεί αν θέλετε, μια τεχνική διαφοροποίηση και ένα διαχωρισμό αυθαίρετο μεταξύ διαφορετικών περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εδαφικέ ανισότητε παρόλα αυτά αυξάνονται και πάρα πολλέ φορέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ, ακόμα και στο πλαίσιο κάποιων χωρών, όπου έχουμε αγροτικές μεγάλες περιφέρειες που θεωρούν ότι μόνο οι ελίτ των πόλεων τελικά υποφελούνται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι η πολιτική συνοχή δεν ξεχνάει κανέναν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες και σε όλες τις γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι συνάδελφοι το λένε αυτό στη γνωμοδότησή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε χρησιμοποίηση όλων των ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη, προκειμένου πραγματικά να μπορούμε να φτάσουμε σε όλε τι περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω των κατάλληλων επενδύσεων να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή. Κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη δέσμευσή σα και νομίζω ότι ε, πραγματικά θα πρέπει να χαιρετήσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προφανώ μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο, αλλά με την οποία συμφωνούμε όσον αφορά τα σημαντικότερα σημεία τη. Ο κύριο Λάντεργκερ τώρα έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, Σήμερα η Επιτροπή των Περιφερειών θα εγκρίνει μια σειρά γνωμοδοτήσεων για την ε, πολιτική συνοχή. Εγώ θέλω να σα ε, δηλώσω τα εξή Ότι υπάρχει μεγάλο βαθμός ε, συμφωνίας, σύγκληση απόψεων, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Οι πόλεις και οι περιφερειέ θέλουν να υπάρχει μια στιβαρή πολιτική συνοχή. Είναι ένα εργαλείο, θα μπορούσαμε να πούμε, για τι επενδύσει, για την ανάπτυξη. Δεν θέλω να προτείνω κάποιες τροποποίησεις για τα όσα έχετε προτείνει. Ε, θα πρέπει όμως να είμαστε ξεκάθαρα στην προσέγγισή μας και επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. Ε, ό,τι, ό,τι αγγίζει εμάς σε τοπικό επίπεδο. Θέλουμε απλούστευση να συνδέονται όλα με τις τοπικές ανάγκες. Επίσης, έχω να σας πω ότι πολλές από τις γνωμοδοτήσεις αυτές ε, βάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά το κλίμα. Αυτό δεν εκπλήσει, αλλά θα πρέπει βέβαια να έχουμε υπόψη το ότι η Συμφωνία των Παρσίων για το κλίμα έχει υποστεί μεγάλα χτυπήματα από τους λαϊκιστές και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού. Αυτό να το εκλάβουμε ως καμπανάκι κινδύνου. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτωπο θα πρέπει να προσέξουμε, θα πρέπει εμείς ως ε, αρχές τοπικές, περιφερειακές να αποσπάσουμε τις επενδύσεις που χρειάζονται για το κλίμα. Παρακαλώ, εγώ μας πάρετε αυτή την υπόθεση πάρα πολύ σοβαρά. Και τώρα κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας πω όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, ιδίω τα Ταμεία και τα Κονδύλια της Συνοχής, να είμαστε συνεπείς, θα πρέπει να πρετανεύει η ισότητα σε κάθε της ε, έκφανση, ιδίω όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων. Αυτό θέλω να σας επισημάνω. Από όπου και αν προέρχονται οι γυναίκες, ό,τι θρησκεία και αν πιστεύουν, υφίστανται δεσμενείς διακρίσεις. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα κονδυλία της συνοχής. Γι' αυτό σας λέω. Να υπάρχει μια πρικοδότηση για την ισότητα και αυτό να συνοδεύσει την ε, πολιτικής συνοχής. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε θα χαθούν πολλές ευκαιρίες για καινοτομία, πολλές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Άρα να μην ξεχνάμε την υπόθεση της όντας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε. Παύλ Μπράντερ. Κυρία Επίτροπε Καρέτσου, Απλώ του ΙΣΙΑΡ χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Τα έχουμε πει τα τελευταία χρόνια συχνά. Αλλά πάντα είναι τιμή μα να βρίσκεστε εδώ. Η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται στις τραπέζι με τις σχετικέ προτάσεις. Τέλειωσε η προπαρασκευή, όλες αυτές οι συζητήσει για την πολιτική συνοχή και μπράβο που μας είχατε ως ισότιμους συνομιλητές και ακούσατε τη φωνή μας σε πολλά θέματα διασυνορικής εργασίας ήμουν εισηγητής όλα αυτά μπήκαν σε κανονισμούς είχατε την ε, γνωμοδότηση ιδιωτικής ε, ε, συγγνώμη, ιδέας πρωτοβουλίας όλα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά για κοινότητες, δήμους και να, αυτό ήταν ακόμα μια έκφραση της καλής ε, συνεργασίας. Τώρα, είμαστε σε άλλη φάση της νομοθετικής διαδικασίας. Ήρθε ένα θέμα ο ρόλος του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Και πάλι θα πρέπει να μας θεωρείτε ισότιμους συνομιλητές. Επίσης και στην προγραμματική διαδικασία και στη φάση της υλοποίησης της πολιτικής αυτής. Να εξασφαλιστεί ότι τελικά οι πόροι θα φτάσουν σε πόλεις, σε περιφέρειες, θα καλύψουν τις τοπικές ανάγκες. Αυτό θα γίνει εάν γίνει σεβαστή η προβλεπόμενη εταιρική συνεργασία. Μισό λεφτάκι μου μένει, οπότε ακούστε κάποιε άλλε προτάσει για το μέλλον. Πρέπει να αλλάξουμε το πώς επικοινωνούμε, πώς ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα. Η προστιθέμενη αξία της πολιτικής είναι ότι φτάνει στο τελευταίο χωριό σας, στην άκρη της περιφέρειας και καλύπτει το, το, τον, τελευταίο, τελευταίο πολίτη, οπότε δεν αρκεί να βάζουμε μία ταμπέλα, μία ευρωπαϊκή κοινοτική σημαία. Θα πρέπει να επενδύουμε στο, ότι βγαίνει από αυτή την πολιτική στην ζωή του κόσμου, του πολίτη. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Νομικτάρση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επίτροπε, μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι η πολιτική αυτή έμεινε στο θεματολόγιο. Εγώ ήμουν εισηγητή για το θεματολόγιο των πόλεων. Ευχαριστούμε γιατί 6% του ERDF πήγε σε επενδύσει όσον αφορά τη βιώσιμη έξοδο των πόλεων και σε σχέση με το, τη σχετική ε, ε, πρωτοβουλία υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να βελτιώσουμε την λειτουργία των πόλεων στο μέλλον. Είναι θέμα που πρέπει στο μέλλον να συζητηθεί να αξιοποιήσουμε την εμπειρία αυτών των ε, εταιρικών σχέσεων, αυτής της συνεργασίας και σε σχέση με τις πολυεπίπεδες δράσεις διακυβέρνησης και να μην έχουμε απλώς κάποιες ασκήσεις ε, δικτύωσης. Να προσπαθήσουμε να βρούμε τις λύσεις για όσους ε, παίρνουν μέρος σε αυτή την υπόθεση. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την υλοποίηση της επικορικότητας. Οι εταιρικέ σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν να έχουμε τις πολιτικές που βελτιώνουν τις πόλεις παντός μεγέθους. Πήγα σε μια διάσκεψη στη Βιέννη για τη στέγαση, σε αυτό το επίπεδο συνεργασία. Πάρα πολύ αξιόλογη με η συνάντηση. Ε, οπότε θα πρέπει να προσέξουμε τι κάνουμε τη δικτύωση με το θεματολόγιό μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την Ήπεθρο με την κατάλληλη χωροταξία. Άρα έτσι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτά τα προγράμματα δράσης. Για πέστε μας, τι λέτε για το θεματολόγιο των ε, πόλεων. Θα προχωρήσει πέρα από τα σχετικά ε, προγράμματα. Μάρκου Μαρκούλα, πρώτος αντιπρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητή Κορίνα, θα ήθελα να τονίσω κάποια σημαντικά κέρια σημεία. Δημιουργούμε τώρα το πλαίσιο για τα τελικά, αν θέλετε, στοιχεία, συστατικά στοιχεία της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής έχει να κάνει με το σχηματισμό. Είναι ένα εργαλείο μεταμόρφωσης πολύ σημαντικό. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει όμως, πέρα από τις διαδικασίες, να ασχολείται και με το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να αποφύγουμε οποιονδήποτε κατακαιρματισμό. Είναι πολύ σημαντικό η πολιτική συνοχή να ενσωματώνει και τη χρησιμοποίηση άλλων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπω για παράδειγμα ορίζοντα 2020, ψηφιακή Ευρώπη και άλλα εργαλεία τα οποία έχουμε ήδη διαθέσιμα. Νομίζω λοιπόν ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να ενσωματωθεί σε τοπικό και, ευρωπαϊκό, και τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με τι δυνατότητε ιδιωτική συγχρηματοδότηση η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις για στοχευμένα μέτρα. Επ' αυτού λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στα διδάγματα τα οποία αντλήσαμε από τη στρατηγική εφιούς εξειδίκευσης. Είδαμε ότι οι περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της στρατηγικής αυτής ήταν σε θέση να συνεργαστούν μεταξύ τους πολύ περισσότερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε στα πλαίσια της συζήτησης τι σημαίνει διασυνοριακό ομόφωνο Επιτροπή των Περιφερειών έχουμε πει ότι προφανώς θα πρέπει και τη χερσαία επικράτεια να λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά και την παράκτια θαλάσσια διάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε στη δική σας συνιστόσα 5 της πολιτικής συνοχής, βλέπουμε αυτήν την διαπεριφερειακή καινοτόμα συνεργασία. Αν η έκβαση τελικά των διαπραγματεύσεων είναι ότι θα εξαφανιστεί η διάσταση αυτή, τότε πραγματικά, κύριε Επίτροπε, φοβάμαι ότι θα χαθεί και ο σχετικό στόχο. Α βρείτε λοιπόν την καλύτερη δυνατή λύση σε σχέση με όλε τι υπόλοιπε συνιστώσει πολιτική συνοχή, ότι η διάσταση αυτή να τηρηθεί. Δηλαδή, οι καινοτόμε, αν θέλετε, περιφέρειε, οι περιφέρειε καπανή, να καταφέρουν να συνεχίσουν το έργο το οποίο ήδη έχουν ξεκινήσει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπου συνεργαζόμενε με τους τοπικά ευθύνοντες, με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο αλλά και με άλλες περιφέρειες μπορούν πραγματικά να πετύχουν πολύ σημαντικούς στόχους όπως και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των εθνών. Τέτοια απτά αποτελέσματα χρειαζόμαστε στο μέλλον και βασίζομαι σε εσά για να πετύχουμε τα θετικά αυτά αποτελέσματα. Πέντε ακόμα συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο. Τονίζω ότι ένα λεπτό χρόνο αγόρευσης έχουμε για τον καθένα. Αλέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλωσορίσατε και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι στόχοι σας και η ε, υπευθυνότητα και οι ευθύνες σας ε, συνάδουν και πολλοί και ταυτίζονται και με τις δικές μας συμφωνώ με τα όσα είπαν ε, η κυρία Μάριν και ο κύριο Σνάιντερ για την διασυνοριακή συνεργασία, την εδαφική συνεργασία ή το δημογραφικό. Τώρα όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάτι που αφορά ιδιαίτερα τη δική μου περιφέρεια που είναι η Γαλλικία στην Ισπανία. Υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες που βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Και υπάρχει το δημογραφικο τωρα ομω θα ηθελα να επικεντρωθω σε κατι που αφορα ιδιαιτερα παράδοξο. και αλλε ευρωπαικε περιφερειες που βρισκονται στην ιδια μοιρα και υπαρχει το γεγονός το γεγονο οτι το ΑΕΠ μα μειώνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, Είμαστε τώρα σε μετάβαση δηλαδή από ανεπτυγμένη περιφέρεια, αλλά η πρικοδότησή μας μειώνεται κατά 40% και ε, περισσότερο, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που λέει το παράρτημα 22 ε, του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Σε τι οφείλεται αυτό εν μέρη ε, στην ειδική μεταχείριση που μας επιφυλάσσει η σημερινή περίοδος. Γιατί για πρώτη φορά περάσαμε από τις λιγότερο ανεπτυγμένες στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Άρα, μιλάμε τώρα για διπλή τιμωρία. Μειώνεται το ΑΕΠ μας κατά 10% και ταυτόχρονα μειώνεται και η πρικοδότηση. Πράγμα που είναι τελείως αντίθετο, θα συμφωνήσετε με το πνεύμα ε, και το στόχο της πολιτικής συνοχής. Άρα, συνεργαζόμαστε με τους βουλευτές για να προσπαθήσουμε να ε, καταφέρουμε καμία περιφέρεια που κατεβαίνει η κατηγορία να μην χάσει Ε, είναι το 1,01 το ΕΠ, το ξέρουμε. Ο χρόνο σα τελείωσε. Ε, η επόμενη συνάδελφο έχει το λόγο. Μπέρκι Τονέιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, και ε, για την παρουσία σας και για την ομιλία σας. Θέλω να σας ε, υποβάλω τέσσερα θέματα. Πρώτον, και για τη δική μου περιφέρεια είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συντελεστές ή χρηματοδότησες να παραμείνουν και σε καμία περίπτωση να μην πέσουν κάτω από το 70% τα είπε ο συνάδελφος Σνάιντερ και σε εμά είναι πάρα πολύ διαφορετική η κατάσταση. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες ίδιες. Δεύτερον, εγώ είμαι ρητά υπέρ του κανόνα νήσιν 3, διότι για τα δικά μας έργα χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό με ασφάλεια και βεβαιότητα βεβαιότητα και έτσι ε, βάζουμε και τα θεμέλια και τα ορόσημα. Χρειαζόμαστε ασφάλεια στον προγραμματισμό. Τρίτο σημείο. Ε, το δικό μου ομόσπονδο κρατήδιο ε, στην τρέχουσα περίοδο έχει ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση από διάφορα ταμεία και το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γιατί δεν είναι μονοδιάστατη ανάπτυξη ούτε τα έργα, είναι διάφορες τομεακές πολιτικές, κλαδικές που συνεργάζονται και σε μια τέτοια ενωμένη περιφερειακή πολιτική θα πρέπει ε, ε, να ε, μπαίνουν και άλλα ταμεία, το είπε και συνάδελφος Μαρίνη. Και το τέταρτο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι οι μειώσεις στα προγράμματα Interreg πρέπει να καταργηθούν. Γιατί το πρόγραμμα Interreg ρίχνει σύνορα, προάγει και την ευρωπαϊκή δουλειά και το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Ευχαριστώ. Επόμενο συνάδελφο. Ε, dear Madam ε, Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον κανονισμό κοινών διατάξεων, τον CPR. Λέει ότι ο ΦΠΑ θα είναι επιλέξιμο κόστος μόνο για σχέδια μέχρι 5 εκατομμύρια. Και λέει ότι αυτό το κατόφλι ως τέτοιο κόστος μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ελκυστικότητας για τους ετούντες, ιδίως για τα έργα υποδομής, γιατί αυτά τα λέει η γνωμοδότησή μας. Το να μην είναι επιλέξιμος αυτός ο ΦΠΑ σε σχέση με χαμηλότερη συγχρηματοδότηση θα κάνει λιγότερο ανταγωνιστική την πολιτική της συνοχής σε σχέση με το ΕΦΣΥ. Και τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Επίσης είναι δυνατόν οι ετούντες να θέλουν να χωρίσουν, να σπάσουν τα έργα. Οπότε για πετε μας, γιατί, ολογική σκέψη το κάνετε αυτό και ποιες θα είναι οι συνέπειες του ότι θέλετε αυτοί οι κανόνες να συνεχίσουν να ισχύουν όσον αφορά τους τωρινούς κανόνες για το ΦΠΑ, τους ω επιλέξιμους. Μικαέλα Φανέλη Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πάλι ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Μαζί κάναμε αυτή την ε, πορεία. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια που έχετε καταβάλει. Φτάσαμε τώρα σε μια αποφασιστική φαστιντηλική ευθεία. Και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε έτσι να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Και αυτό γιατί βλέπετε όμως ότι έχουμε ομοφωνία στην Επιτροπή των Περιφερειών για την έγκριση αυτών των ε, γνωμοδοτήσεων γιατί είναι πολύ σπουδαία τα αποτελέσματα σωστή συμβουλή και γι' αυτό και εμείς επιδοκιμάζουμε την ουσία του περιεχομένου. Περισσότερη συνοχή για τις πόλεις και για την Ήπεθρο. Αυτό θέλω να αναδείξω το θεματολόγιο της ε, πόλης που τονίστηκε από έναν προελίσσαντα συνάδελφο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο το ε, δοκιμάσαμε και το οποίο ε, ενισχύθηκε κυρίως όσον αφορά το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου. Είναι πολύ σημαντικό ορόσημο. Έχετε περάσει το χρόνο αγόρευσης, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Αγοραστός έχει το λόγο. Άρα θα, αυτό θα πρέπει να περιβάλλουμε την, ε, το θέμα την Ήπεθρο. Κύριος Αγοραστός. Επίτροπος, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πραγματικά δημιουργικές υπηρεσίες τις οποίες προσφέρατε. Με ταχύτητα, δημιουργικότητα, συνεργασία και συνέργεια καταφέραμε πάρα πολλά να επιτύχουμε και μάλιστα να κάνουμε και πράγματα τα οποία φανταζόταν αδύνατα στο παρελθόν. Κυρίε και κύριοι, το... η νέα πολιτική συνοχής πρέπει να είναι γρήγορη εφαρμόσιμη συνεργατική αποτελεσματική και θα πρέπει να προεξοφλεί το μέλλον και όχι να μελοποιεί το παρόν. και βέβαια χρειάζονται τέτοιες πολιτικές ούτως ώστε να χτυπηθεί η γραφειοκρατία η κακονομία η πολυνομία και οπωσδήποτε να δώσει μια ταχύτητα γιατί ο χρόνος είναι θέσεις εργασίας που λείπουν από την ευρώπη είναι χρήμα στην πραγματική οικονομία που λείπει από την πραγματική οικονομία της ευρώπης. για να πετύχουμε πρέπει να ακολουθήσουμε το μότο be the change you wish to see in the europe. Thank you. Euh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Σας ζητώ συγγνώμη ήμουν τόσο αυστηρός με το χρόνο αγόρευσης. Δεν είχα άλλη επιλογή. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να εξασκηθούμε αρκετά προκειμένου να μπορούμε να τηρούμε το χρόνο αγόρευση. Χωρί περαιτέρω καθυστέρηση δίνω το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει σε όλε αυτέ τι παρατηρήσει και τι ερωτήσει που ακούσαμε από του συναδέλφου. Σα ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τα μέλη τη Επιτροπή των Περιφερειών. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι άκουσα τι παρατηρήσει αυτέ. Ξέρετε ότι είχαμε όλε αυτέ τι συνεχείς συζητήσεις τα τελευταία αυτά χρόνια και γνωρίζω ότι άλληλο υποστηριχθήκαμε όσον αφορά την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, αλλά είχαμε και διαφορετικές προσεγγίσεις ε, σε άλλα σημεία. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω σε κάποια από τα σημεία τα οποία θίξατε και θα προσπαθήσω έτσι να εξηγήσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία υποβλήθηκε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 2 Μαΐου του 2018. Τονίζω όμως ευθύ εξ αρχής ότι η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται πλέον στα χέρια των συνομοθετών, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο δηλαδή. Αν θέλετε όμως εσείς να αλλάξετε τώρα κάποια στοιχεία της πρότασης αυτής, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με τα κράτη-μέλη, με τις κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη σας, με τους προέδρους, πρωθυπουργού που εκπροσωπούν τη χώρα σας στο Συμβούλιο. Θα γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη στα δύο αυτά θεσμικά όργανα. Την προηγούμενη Παρασκευή είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τους υπεύθυνους για την περιφερειακή πολιτική από τα κράτη-μέλη. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι διεξάγεται μια συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βέβαια στηρίζομαι σε εσά προκειμένου να έχουμε θετικέ γνωμοδοτήσει τη Επιτροπή των Περιφερειών, ευνοϊκέ για την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέρουσε ε, σωστά επιχειρήματα και ξέρετε ότι εγώ ανέκαθεν εκτιμούσα πάρα πολύ τη μεταξύ μου συνεργασία. Θα απαντήσω στα ερωτήματά σας ένα προς ένα όσον αφορά τον προγραμματισμό 5 συν 2. Νομίζω ότι δεν απέχουμε τελικά πάρα πολύ στι προσεγγίσεις μας. Ξέρω ότι εσείς έχετε ακόμα κάποιους ενδιασμούς. Παρ' όλα αυτά ξέρω ότι επί της αρχής υποστηρίζετε την αρχή της ευελιξίας και εσείς, προκειμένου να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε νέες αναδυόμενες καταστάσεις. Ας δούμε λοιπόν πώς η αρχή αυτή της ευελιξίας θα εφαρμοστεί στην πράξη. Όπως σας είπα, η πρότασή μας προβλέπει και τη δυνατότητα αναθεώρησης και συνέχειας. Στόχος μας δεν είναι να ξεκινήσουμε από το μηδέν μετά από πέντε χρόνια, όπως είπε ο κύριος Σνάιντερ. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε έργα τα οποία ακολουθούν διαφορετικές προγραμματικές περιόδους, αλλά αν τροποποιηθούν τελικά οι ανάγκες ή αν δούμε ότι δεν μπορούμε τελικά μέσα σε πέντε χρόνια να δαπανίσουμε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να διευκολύνουμε τη μεταφορά κονδυλίων από τον έναν άξονα στον άλλον. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε την αρχή 5 συν 2. Όσον αφορά την προχρηματοδότηση και την συγχρηματοδότηση, καταγράφω τι ανησυχίε για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει να σας πω ότι ε, πιστεύω ότι η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά ρεαλιστική, γιατί στην πράξη θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση ακόμα και με μειωμένο προπολογισμό. Κατά την άποψή μας, η αύξηση της χρηματοδότησης δημιουργεί μεγαλύτερο βαθμό ενστερνισμού επιτόπου και η πρόταση λοιπόν χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι κάτι το νέο, Ουσιαστικά θέλουμε να επιστρέψουμε στα επίπεδα προ-κρίσης, όταν είχαμε δηλαδή άλλα τότε επίπεδα σε χρηματοδότηση. Αυτά λάβαμε υπόψη μας και θεωρήσαμε ότι με τον μειωμένο υφιστάμενο προπολογισμό μετά από κάποια χρόνια οικονομικής ανάπτυξης θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε κάποια στιγμή στα επίπεδα πρώτης κρίσης. Βλέπω όμως ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ίδια στάση με εσά. Υπάρχει μια κάποια αντίδραση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όσον αφορά τον ε, θεματικό, τη θεματική συγκέντρωση. Ξέρετε ότι ε, πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες προτεραιότητες. Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, αναγκαστικά θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, ιδίω ε, για την μορφή που θα πάρει η οικονομία στο μέλλον. Πρέπει να επικεντρωθούμε και σε άλλους τομείς όπως το περιβάλλον, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια ε, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε μια νέα ανακοίνωση όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προτείνουμε λοιπόν μέσω της θεματικής συγκέντρωσης ένα ευέλικτο σύστημα. Έχουμε πιο ευρείες κατηγορίες πλέον από ό,τι στο παρελθόν και να πόκειται πλέον στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες να καθορίσουν τις κατηγορίες αυτές. Είναι πιο εύκολο, με άλλα λόγια, να μετακινήσει κανείς ε, τη χρηματοδότηση από τον έναν κλάδο στον άλλον. Και κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε και μια μεγαλύτερη γκάμα θεμάτων, περισσότερες προτεραιότητες. Όσον αφορά τώρα το 1 συν 2, καταγράφω τις ανησυχίες σας. Πάλι εδώ πέρα το μέτρο απλούστευσης το οποίο εγκρίναμε θεωρούμε ότι θα επιταχύνει την υλοποίηση και την εφαρμογή. Έντονα επικριτική ήταν η στάση όσον αφορά τις ε, καθυστερήσεις. Θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να απλουστευτεί περισσότερο το σύστημα όσον αφορά την επιλογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και πώ αυτά θα χρηματοδοτούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με την πρόταση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και με την αρχή νήσιν 2 αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα. Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στο νήσιν 2 και αυτό χάρη στην προβλεπόμενη απλούστευση και θεωρώ ότι η επιστροφή στην αρχή νήσιν 2 θα λειτουργήσει πολύ θετικά και για τη φήμη την υπόλοιψη της πολιτικής ε, συνοχής. Όσον αφορά τώρα το ίντερεγκ. Συμφωνώ μαζί σας, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει, αφορά περίπου 30 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι ζουν σε παραμεθόριες περιοχές. Εγώ είμαι σαφώ υπέρ αυτή της διασνοριακής συνεργασίας. Από κοινού με τον Καρλ Χάινς επισκέφθηκα την δικιά του περιοχή, που ουσιαστικά έχουμε μια παραμεθόριο περιοχή που αφορά όχι μόνο δύο, αλλά τρεις χώρες, είναι πολύ σημαντική λοιπόν εκεί η προβλεπόμενη συνεργασία και με τον πρόεδρο της Περιφέρειας των Αζωρών είχα τη δυνατότητα να συζητήσω περισσότερο αυτά τα οποία είπατε και την προηγούμενη εβδομάδα στις Κανάριες νήσους, όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παράκτιες περιοχές και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι ιδιαίτερα απόκεντρε περιφέρειε. Πρέπει εδώ να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα δεσμευμένη όσον αφορά την θαλάσσια συνεργασία, συνεργασία μεταξύ παράκτιων περιοχών. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα ζητήματα που θίξατε, η αστική διάσταση. Θα γνωρίζετε ότι ο κανονισμό περί κοινών διατάξεων προβλέπει μια συγκεκριμένη πλέον πολιτική προκειμένου οι πολίτε να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσοντα περισσότερο τι αστικέ υπαίθριε και παράκτιες περιοχές, προκειμένου να υπάρχει μια πολυτομιακή προσέγγιση για την ανάπτυξη. Και εκεί έχουμε και συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά τις πόλεις. Ένα τουλάχιστον 6% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ προβλέπονται για έργα τα οποία αφορούν πόλεις και αστικά κέντρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά να επιτρέψουμε στους δημάρχους των πόλεων, να σχεδιάσουν τη δική του στρατηγική. Γιατί εσεί γνωρίζετε πολύ καλύτερα από ότι εμεί στι Βρυξέλλε ποιε είναι οι ανάγκε σα. Εσεί στι μεγάλε πόλει, στι πρωτεύουσε, ξέρετε τι χρειάζεται και ξέρετε τι είναι περιττό. Τώρα, για να ανταποκριθώ περισσότερο, να απαντήσω μάλλον στην ερώτηση που ακούστηκε για την ε, αστική πρωτοβουλία. Στα πλαίσια τη αστική πρωτοβουλία έχουμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση για όλε τι πόλει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συσπηρώνονται σε ένα κοινό πρόγραμμα όλα τα αστικά εργαλεία τα οποία είχαμε στο παρελθόν μέσω κοινή διαχείριση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θα θέλαμε να συσπηρώσουμε και να ομαδοποιήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα, Urban, Urbact, προγράμματα ανάπτυξης των πόλεων, δίκτυα διαβίβαση τεχνολογιών και γνώσεων, καθώς επίσης και όλους τους υπόλοιπου μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με την αστική πολιτική. Θα βρισκόμαστε εδώ πέρα σε καθεστώ έμεση συνεργασία, όπω είχε συμβεί στο παρελθόν με τέτοιε αστικέ πρωτοβουλίε. Και αυτό που θέλω να πω προ όλου είναι ότι είμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε. Είμαστε στη διάθεσή σα για να σα δώσουμε περισσότερε καθοδηγήσει, Θεωρώ πάντω ότι αυτή τη στιγμή με τη νέα αυτή προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφεύγουμε πλέον τον κατακαιρματισμό που είχαμε στο παρελθόν όσον αφορά τι αστικέ πρωτοβουλίε. Όσον αφορά τώρα το φόρο τη θέμενη αξία, οι σχετικέ διατάξει για την περίοδο 2014-2020 οδήγησαν σε ανασφάλεια δικαίου, σε νομική αβεβαιότητα και σε προβλήματα για πάρα πολλέ τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Οι διατάξει αυτέ αναφερόντουσαν στου εθνικού κανόνε φόρου προστιθέμενη αξία και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν πάρα πολλές ε, διαφορές και ανισότητες μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών στο πλαίσιο των κρατών μελών. Προκειμένου να πλουστεύσουμε τα πράγματα για τις ε, αρχές προγραμματισμού και για τους δικαιούχους ε, προβλέπουμε έναν απλό κανόνα για τα έργα που είναι κάτω των 5 εκατομμυρίων επιλέξιμος φόρος προστέμενης αξίας αυτόματα, ενώ δεν θα είναι επιλέξιμος ο φόρος προστέμενης αξίας για τα έργα πάνω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα εξαρτάται πλέον το κριτήριο αυτό από τα εθνικά κριτήρια, από τον εθνικό φόρο προστέμενης αξίας. Βλέπουμε επίση ότι τα περισσότερα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ή βρίσκονται κάτω του κατοφλίου αυτού των 5 εκατομμυρίων, άρα δεν πρόκειται να ζημιωθούν οι δικαιούχοι. Επίση όσον αφορά πάντα το φόρο τη αξίας, θα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε περισσότερα προγράμματα στο μέλλον, διασφαλίζοντας και τον προπολογισμό όμως της πολιτικής συνοχής για τα επόμενα χρόνια, όσον αφορά το ζήτημα της ισότητας των φύλων. Ζήτημα ιδιαίτερα προσφυλές για μένα. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα θετικό ότι στα πλαίσια του κανονισμού περί κοινών διατάξεων τίθεται πλέον και το ζήτημα της μη εισαγωγής διακριτικής μεταχείρισης, το ζήτημα της ισότητας των φύλων και της ισότιμης μεταχείρισης. Είναι σημαντικό το ότι γίνεται πλέον συγκεκριμένη αναφορά. Στην πράξη όμως οι αρχές αυτές θα πρέπει να τηρούνται καθότι ούτω ή άλλω ανήκουν στο κοινοτικό κεκτημένο και ουσιαστικά είναι αρχέ που θα πρέπει να διέπουν τη στάση όλων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αρχέ που άλλωστε προασπίζονται και στα πλαίσια του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό εκ των προτέρων και προληπτικά να θέσουμε τη διάσταση αυτή, να αποτελεί προτεραιότητα και σε εταιρικέ σχέσεις και στα μελλοντικά έργα τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν αντί να έρθουμε εκ των υστέρων να θεραπεύσουμε τα κακό, σκήνεμα, τα κακό σκήμενα. Επίσης, ήδη αρχής γενομένης από του χρόνου, ακριβώς επειδή έχουμε και πάρα πολλές εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές τοπικές εκλογές, είναι πολύ σημαντικό να διεξιάγουμε και μία εκστρατεία για περισσότερες γυναίκες στην δημόσια διοίκηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε οι οποίε διστάζουν τελικά να θέσουν αυτούς υποψήφιες στις δημοτικές εκλογές για τη θέση του Δημάρχου ή για να συμμετέχουν σε δημοτικά συμβούλια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήδη από το 2019 θα πρέπει να ξεκινήσει και μια πιο ενεργή εκστρατεία προκειμένου να έχουμε υψηλότερη συμμετοχή γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όσον αφορά το Brexit, ξέρετε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει πλέον ένα σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης. Περιμένουμε όμως τώρα και την απόφαση του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Θλιβερή κατάσταση βέβαια που αντιμετωπίζουμε. Είχαμε μία πρόταση το 1975, η οποία επιβλήθηκε ουσιαστικά από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, όταν χρειάστηκε τότε να κλείσουν πάρα πολλά ορυχεία, θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε την πολιτική συνοχή με 27 κράτη-μέλη. Ας δούμε όμως ποια θα είναι η απόφαση στις 11 Δεκεμβρίου από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Κάποιες τελικές παρατηρήσεις πρέπει να σας πω ότι πάντα αφουγκράζομαι τις ανησυχίες σας. Είμαστε εδώ πέρα όλοι φίλοι της πολιτικής συνοχής και εμβαθύνουμε εμεί ακόμα περισσότερο στι ανησυχίε σα για να δούμε τελικά πώ θα προσαρμόσουμε του πόρου μα, ποιε νέε δυνατότητε μα δίνονται και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι είστε στο πλευρό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη διαδικασία πλούστευση. Γιατί ξέρετε ότι για τέσσερα ολόκληρα χρόνια ακούω παντού τι ανησυχίε, οπουδήποτε και πηγαίνω, γραφειοκρατία, πολύπλοκε διαδικασίε. Πάνω από 80 μέτρα απλούστευση προβλέπονται στη νέα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι πάρα πολύ που τα υποστηρίζετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να μα υποστηρίξουν και τα κράτη-μέλη, έτσι δεν είναι. Γιατί αν εμεί έλθουμε και απλουστεύσουμε του ε, βασικού κανονισμού που ε, αποτελούν ουσιαστικά και το ίμιση τελικά των συνολικών κανονισμών που έχουμε και αν παράλληλα τα κράτη-μέλη δεν μας ακολουθήσουν και από τη δικιά τους την πλευρά έρθουν να δημιουργήσουν περισσότερες κανονισμούς και περισσότερες διαδικασίες, δεν πετυχαίνουμε τίποτα στην πράξη. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που διατηρείται φιλική, διάστηση, φιλική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνούμε για τα περισσότερα ζητήματα από ό,τι βλέπω. Για κάποια άλλα ζητήματα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης, όπως είπατε. Από την άλλη όμως το περιθώριο ευελιξίας που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλο, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνω κάθε ό,τι μπορώ, προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο σε μια κοινή απόφαση. Ξέρετε ότι ελπίζω ότι στο πλαίσιο του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και με την Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε θετικές αποφάσεις, να μπορέσουμε δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του 2019 να δρομολογήσουμε όλα τα προγράμματα. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν αντλήσει θετικά διδάγματα από το παρελθόν όλα τα κράτη-μέλη και πολύ φοβάμαι ότι αν καθυστερήσουμε και αν περιμένουμε πρώτα να διεξαχθούν οι ευρωεκλογέ, θα καθυστερήσουμε την έγκριση τη νομοθεσία και θα καθυστερήσουμε τη συνεχεία και την έναρξη των προγραμμάτων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από κοινού να δώσουμε μια κοινή μάχη και να έχουμε μια τελική συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ για τις γνωμοδοτήσεις αυτές. Συγχαίρω όλους τους εισηγητές. Σας είμαι πραγματικά ευγνώμων, γιατί κι εσείς δίνετε μια σημαντική μάχη για μια πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, για σημαντικές οικονομικές προοπτικές, για δυνατότητες εξυγχρονισμού των περιφερειών, για τη δυνατότητα εφαρμογής οικολογικών πολιτικών, για περιφέρειες οι οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν πιο ομαλά όλες αυτές τις νέες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς και ας δούμε πώς θα διεξαχθούν τα πράγματα στο τέλος της εντολής μας. Νομίζω ότι ήταν ε, η τελευταία φορά που σας είδα τουλάχιστον για το 2018. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές διακοπές σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και για σας και για τις οικογένειές σας και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλατε προκειμένου να βελτιώσουμε τις ζωές των πολιτών μας στις περιφέρειές μας, στις πόλεις μας και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ορίστε, πολύ ωραία συζήτηση αυτή εισαγωγική για τις συζητήσεις. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα έτσι ώστε μετά τις γιορτές ε, να προχωρήσουμε και σας ευχόμαστε και εμείς ό,τι το καλύτερο. Και να πούμε στην τελική ευθεία και να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που από κοινού ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη. Επανέρχομαι στις ανακοινώσει βέβαια, για να σας πω τα εξή. Η έκδοση 2020 του βραβείου ε, και, ε, καινοτόμα ε, ε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε στις 19 Νοεμβρίου ε, στο Γκράτς της Αυστρίας στην αντίστοιχη ε, διάσκεψη. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα σήμα αριστεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινοτομία, για την πρόθεση της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού κλίματος. Και βραβεύει ε, ακριβώς ε, τις πιο πιστικές προσπάθειες και δίνει και μεγάλη προβολή ε, στην περιφέρεια που παίρνει το βραβείο. Σας ευχαρίνω να καταθέσετε υποψηφιότητα για το σήμα αυτό επιχειρηματικότητας. Επιτρέψτε μου επίσης να σας θυμίσω ότι αυτό δεν απευθύνεται μόνο στις περιφέρειες, αλλά και στις διασυνοριακές περιφέρειες και στους δήμους και τις κοινότητες. Υπάρχει προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 27 Μαρτίου 2019 και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες ε, σε ένα σταν περίπτερο εδώ ενημερωτικό στην ε, έξοδο της αίθουσας. Θα βρείτε επίσης το χρονοδιάγραμμα των ε, συνεδριάσεων μας για το 2019. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στις εξης ημερομηνιε ημερομηνίες 14-15 Μαρτίου όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής ε, των Περιφερειών και των Δήμων ε, στο Βουκουρέστι. Σημειώστε παρακαλώ από τώρα αυτή την ημερομηνία, 14-15 Μαρτίου. Και επίσης θα βρείτε στους φακέλους σας δύο έγγραφα που έχουν σχέση με ε, την πληροφορική. Το πρώτο είναι ένα ερωτηματολόγιο για την ικανοποίηση ε, των αναγκών σας και στη συνέχεια οι ε, αντίστοιχε επιτροπές θα το συζητήσουν. Επιτροπή Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων δηλαδή για να βελτιώσουμε τους υπολογιστές μας. Και επίσης θα βρείτε και ένα φυλάδιο ενημερωτικό για την εφαρμογή κύκλος ε, που θα διευκολύνει τη δική σας επικοινωνία με τη γραμματεία μας. Αυτές ήταν λοιπόν οι ανακοινώσεις που ήθελα να προσθέσω στις προηγούμενες που σας εκφώνησα και τώρα νομίζω έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στο κυρίως πιάτο. Τελειώσαμε το απεριτίφ, τελειώσαμε το ορντεύρ, πάμε στο ψητό τώρα. Έχουμε πάρα πολλές νομοδοτήσεις να ε, ε, εγκρίνουμε και αρχίζουμε αμέσως με ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων. Παρακαλώ τους εισηγητές μας, Κατιού Σαμαρίνη και Μιχαήλ Σνάιντερ, να έρθουν εδώ στο Προεδρείο για να μπορέσουμε αμέσως να πούμε στην ουσία των συζητήσεών μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω βέβαια όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπόνηση της γνωμοδότησης αυτής και καταρχάς βέβαια τον συνεισηγητή, τον κύριο Σνάιντερ. Είχαμε μία εξαιρετική επικοδομητική συνεργασία τους τελευταίους αυτούς μήνες και να ευχαριστήσω βέβαια και τους εμπειρογνώμονές μας Καπορίτσι και Φένερ. Να ευχαριστήσω όμως και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικής Εδαφικής Συνοχής και Προπολογισμού, ΚΟΤΕΡ, γιατί χάρη στη συμμετοχή όλων των συναδέλφων καταφέραμε να εκπονήσουμε τη γνωμοδότηση αυτή που σας, που παρουσιάζουμε σήμερα, μια γνωμοδότηση που θεωρώ ότι πραγματικά ανταποκρίνεται στην κοινή θέση όλων των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών. Πιο συγκεκριμένα, θεωρώ ότι η γνωμοδότηση αυτή δεν δείχνει μόνο ότι μάλλον η στάση που κρατά απέναντι στην γνωμοδότηση αυτή δεν δείχνει μόνο την εμπιστοσύνη που έχετε προ εμά, αλλά και την εμπιστοσύνη που έχετε προ το περιεχόμενο τη γνωμοδότηση αυτή, που θεωρώ ότι είναι μια γνωμοδότηση ορόσημο όσον αφορά την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Του τελευταίου αυτού μήνε προσπαθήσαμε πραγματικά να προωθήσουμε το βασικό περιεχόμενο και του βασικού στόχου, τη δεγόμενη συμμαχία, τη συνοχή, όπου όπω σα είπα, απότερο στόχο τη είναι να καλυφθούν όλε οι περιφέρειες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το οποίο τονίζουμε επίση στη γνωμοδότηση αυτή, είναι ότι στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου και στο πλαίσιο των πολιτικών πρωτοβουλειών θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην νέα της ανακοίνωση. Δηλαδή ότι θα πρέπει η πολιτική συνοχή να είναι πιο προβεβλημένη, πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Αν έχουμε κάτι να πούμε προς τους πολίτες μας, αν θέλουμε όντως να τους δείξουμε έναν τομέα όπου η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απτή και θετική, ε, ο τομέας αυτός είναι η πολιτική συνοχής και τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής. Το σχέδιο λοιπόν αυτό της γνωμοδότησης έχει 78 τροπολογίες. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε 32 συγκεκριμένες πολιτικές συστάσεις. Τονίζουμε καταρχάς κάποια κοινά σημεία, δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική συνοχή για όλες τις περιφέρειες, μια αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής που να βασίζεται στις τρεις τρεις μορφές διαφορετικών περιφερειών. Έχουμε επίσης όμως και κάποιες ανησυχίες που ελπίζουμε να εισακουστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες, ιδίως όσον αφορά τον αποκλεισμό, την εξαίρεση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και λέμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε αυτή την ευκταία ολοκληρωμένη σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τα εργαλεία πολιτικής συνοχής και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η νέα του μορφή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχή. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα σημεία που μα ενδιαφέρουν όλου ιδιαίτερω. Το να μπορούμε ως περιφέρειες να καινοτομούμε και να δημιουργούμε και νέες στρατηγικές για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους που να προωθούν την οικονομική βιωσιμότητα. Επίσης, αναφερόμαστε πάρα πολύ στο ζήτημα της απλούστευση. Κάποιε ανησυχίε μα έχουν εισακωστεί. Σε κάποια άλλα σημεία λέμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Σε κάθε περίπτωση, ο απότερο στόχο είναι να μετριαστεί το γραφειοκρατικό άκτο που επιβαρύνει τόσο πολύ το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και πεποδίζει πάρα πολλού πολίτε από ότι έχουν πρόσβαση στα κονδύλια. Λέμε επίση στην πρότασή μα αυτή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε την επανεισαγωγή του κανόνα νήσιν 2. Λέμε ότι θέλουμε τον κανόνα νήσιν 3 και κατά αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να μειώσουμε το οικονομικό κόστος για το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και λέμε ότι στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου θέλουμε κάτι που το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ως Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα για την πολιτική συνοχής να μην συμπεριλαμβάνεται. Εμείς είμαστε κατά της αιρεσιμότητος αυτής Λέμε ανταυτού ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η εταιρική σχέση να λειτουργεί πλήρως ακόμα και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η εταιρική σχέση δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοπικού και περιφερειακού επίπεδου. Προσπαθήσαμε επίσης ε, να συγκεράσουμε όλες αυτές τις προτάσεις και ανησυχίες που ακούστηκαν από όλους τους συναδέλφους και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε και ιδίω τις πολιτικές αυτές συστάσεις προβάλλουμε περισσότερο την πολιτική οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Απόψει δηλαδή που ακούστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια τη τελευταία αυτή θητεία, οι περισσότερε έχουν ω στόχο να βελτιώσουμε την υφιστάμενη πολιτική συνοχή και να καταφέρουμε τελικά να προασπίσουμε περισσότερο το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής. Να καταφέρουμε δηλαδή να συμμετέχουμε κι εμείς όλο, όλο, όσο δυνατόν περισσότερο στην εκπόνηση της πολιτικής συνοχής και στην κατάρτιση των στόχων της πολιτικής αυτής. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής που συμμετείχαν στο εγχείρημα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριο Σνάιντερ, ο συνεισηγητής του Εκτολόγου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την προλαλή σα. Ευχαριστώ κυρία Μαρίνη. Συμφωνώ με όλες τις ευχαριστίες που απευθύνατε στους εμπειρογνώμονες, στη γραμματεία, του συναδέλφους που κάθεσαν τροπολογίες. Συμφωνώ και επί της ουσίας με όλα όσα είπατε και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω συνεπώς. Είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα που από κοινού έχουμε προωθήσει. Αυτό που έχει σημασία τώρα ποιο είναι. Είμαστε κάπως ικανοποιημένοι με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, αλλά έχουμε ακόμα και κάποιες επιθυμίες και προτάσεις για πολύ σαφείς και συγκεκριμένες, που δεν είμαστε ικανοποιημένοι και δεν μας βοήθησε να προχωρήσουμε η σημερινή συζήτηση με την κυρία Κρέτσου, δεν αποκόμισα την αίσθηση ότι μα έκανε και τρομέρε παραχωρήσει, αλλά βέβαια μα είπε ότι δεν έχει τώρα την ηγεσία των διαπραγματεύσεων. Έχει δίκιο. Ε, η υπόθεση είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εμεί λοιπόν με τι προτάσει μα πρέπει να αποταθούμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ωραία. Ε, το καλό ποιο είναι. Το Κοινοβούλιο ανέβαλε την απόφαση του για τους κανονισμούς για τα διορθωτικά ταμεία. Δεν θα αποφασίσει το Δεκέμβριο όπως είχε ε, προγραμματιστεί, αλλά τον Ιανουάριο θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή. Οι δικέ μα 200 τροπολογίες είναι ψηλοπράγματα. Στο Κοινοβούλιο είναι πάνω από 3.000 οι τροπολογίε. Η αρμόδια επιτροπή το συζητάει λοιπόν το Γενάρη και τον Απρίλιο θα πάει στην Ολομέλεια. Έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε με του βουλευτέ μα. Τα σημαντικότερα, νήσιν 2 ή νήσιν 3. Εμεί ξεκάθαρα ε, είπαμε ότι είμαστε κατά του νήσιν 2 και υπέρ του νήσιν 3. Συγχρηματοδότηση. Ε, είμαστε σαφώ κατά τη μείωση των συντελεστών πόρων χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Μιλάμε για 70% για τι περιφέρειες σε μετάβαση. Και τα δύο τα συνοψίζω. Για ποιο λόγο θα θέλουμε όλα αυτά. Διότι η πολιτική συνοχή και τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να μπορούν να δουλεύουν αποτελεσματικά και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Αν μειώσει την περίοδο τη χρονική και αν μειώσει και τη συγχρηματοδότηση, ε, δημιουργεί τι προποθέσει να υπονομευτεί η επιτυχία ε, των ταμείων και να υπολείπεται της ε, τωρινή προγραμματική περίοδου που έτσι κι αλλιώ έχουμε προβλήματα. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, ε, δημιουργούμε τα προβλήματα για την επόμενη περίοδο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτό για μα. Και μετά υπάρχει και ένα θέμα της ευρύ, του ε, εκτός από το ΑΕΠ θέλουμε και άλλους δείκτες. Και η συνάδελφος Μαρίνη συμμετείχε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Μας λείπει λοιπόν όμως και το στοιχείο το δημογραφικό. Σε πολλές περιφέρειες έχουμε πρόβλημα δημογραφικό και τα δημογραφικά προβλήματα είναι εμπόδιο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αλλά και εμπόδιο στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Ακριβώς αυτό που υποτίθεται ότι θα πρέπει να βελτιώσουν τα διευθυντικά ταμεία. Είναι παράλογο να μην λαμβάνονται υπόψη τα δημογραφικά προβλήματα στην κατανομή των πόρων. Ε, είναι στην κεντρική ιδέα, στον πυρήνα της ίδια της λογικής παρέμβασης των διαθροτικών ταμείων. Γι' αυτό ζητούμε να διορθωθεί αυτό, να βελτιωθεί. Επόμενο θέμα, η απλούστευση. Ε, ομολογώ και παραδέχομαι ότι έχει κάνει καλές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διοικητική απλούστευση, για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Εν μέρη βοηθήσαμε κι εμεί με την Task Force και έπιασε τόπο. Το Μάρτιο κάναμε προτάσεις για την απλούστευση της διοίκησης και το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε τις σχετικές αποφάσεις και έλαβε μερικά πράγματα υπόψη. Αλλά όχι μέχρι εκεί που θα θέλαμε. Στην κοινή μας γνωμοδότηση έχουμε συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που μας έρχονται από ανθρώπους που τα εφαρμόζουν στην πράξη, όχι από πολιτικούς, για το πώς μπορεί να απλουστευτεί ακόμα περισσότερο η διοίκηση και να μειωθεί η γραφειοκρατία. Τώρα τι ακούω από τους πρώτους γύρους ε, των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα, ότι ιδιαίτερα από τα κράτη-μέλη έρχονται διάφορες προτάσεις για λεπτομερείς ρυθμίσεις που θα πρέπει λέει, να ε, υιοθετηθούν και να ενταχθούν στον κανονισμό. Εκεί που μειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνονται οι προσπάθειες να ε, μπουν περισσότερες διατάξεις από την πίσω πόρτα. Ε, αυτός είναι ο λάθος δρόμος. Ακριβώς αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε. Περισσότερη μείωση της γραφειοκρατίας και περισσότερη απλούστευση. Αλλιώς ε, υπάρχει κίνδυνο στις διαπραγματεύσεις να πολλαπλασιαστούν αντί να μειωθούν. Και έχουμε και άλλο πρόβλημα να χαθούν επενδύσεις γιατί χάνεται το κόσμο στο χαρτοβασίλειο, ε, στο να συμπληρώνει έντυπα και να μην καταλαβαίνει τις διατάξεις. Αυτά είναι τα σημαντικά ε, θέματα που θα πρέπει να ε, τα λύσουμε συνομιλώντας με τους βουλευτές μας, με τα μέλη των κυβερνήσεων, για να έχουμε καλύτερα διαστατικά ταμεία την επόμενη περίοδο. Και όλα τα πράγματα αυτά θα είναι πολύ πιο δύσκολα αν δεν εγκριθεί εγκαίρως στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αντίστοιχα ο κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία στη συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλες μας τις επαφές και να το προωθήσουμε. Εδώ ομολογώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός. Γενικά σας ευχαριστώ όλους. Κάναμε καταπληκτική δουλειά και αν σήμερα ε, με μια ισχυρή βρόντερη ψηφοφορία ε, το περάσουμε, αυτό θα εντυπωσιάσει και τα άλλα θεσμικά όργανα, γιατί θα πούμε ότι είμαστε συμπαγεί και ενωμένοι, όλη η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άλλο θέλει να πάρει το λόγο στη γενική συζήτηση για αυτό το θέμα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η γενική συζήτηση έγινε παρουσία της κυρίας Επιτρόπου. Νομίζω ότι συμφωνείτε με τη σοφία αυτή που σας είπα. Πάμε στις τροπολογίες. Τρεις είναι. Η πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τρία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία υπέρ της νομοδότησης. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση ομόφωνα. Και συγχαρητήρια στους συγγητές μας για το έργο τους. <laughs> το παρελθόν και το μέλλον. Ε, πάμε στο σημείο 6 την ημερήσια διάταξη. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και ο σχετικός κανονισμός. Θα παρακαλέσω την εισηγήτρια. Μάλλον απουσιάζει η συγκήτρια κυρία Σουζάνα Ντίας Πατσέκο και παρακαλώ τον συνάδελφο που την αντικαθιστά να έρθει να μας παρουσιάσει την γνωμοδότηση. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, σας τα λέω ε, από τι τη τη ε, εισηγήτρης Δίας Πασέκου που δεν μπόρεσε αν και θα ήθελε να βρίσκεται εδώ. Είναι τιμή μα να ολοκληρώνουμε αυτό το οποίο όλοι μαζί το κάναμε και σε στενή επαφή με την Επιτροπή, τις πολιτικές ομάδες και τους εμπλεκομένους. Αυτό το νομοθέτημα για το ΕΚΤΑΦΣΥΝ είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό για μας, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης, γιατί το Ταμείο αυτό υπήρξε και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα της Ένωσης, ούτως ώστε να επενδύει στα πρόσωπα, στον άνθρωπο, και είχαμε τον Οκτώβριο το σχέδιο του νομοθετήματος και εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία. Το σχέδιο νομοδότησης, το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε, περιέχει 46 συστάσεις νομοθετικών τροπολογιών όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε και 32 παραγράφους με πολιτικές συστάσεις. Θα πρέπει τώρα να αναδείξουμε τα πιο σημαντικά μηνύματα γύρω από τα οποία στρέφεται μάλλον αυτό το σχέδιο κειμένου. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαίο οι στόχοι γνωστοί σε όλους, οι παραδοσιακοί στόχοι του ΕΚΤΑΦ για την αγορά απασχόληση, την παιδεία και την κατάρτιση να συμπληρωθούν με νέους στόχους για τους μετανάστες, την υγεία, τους ε, νέους και καταπολέμηση της φτώχειας. Παρ' όλα αυτά, στο σχέδιο κειμένου λέμε ότι ανησυχούμε γιατί ίσως υπάρχει μείωση της προοικοδότησης λόγω της καινούρια κατάστασης το ότι δίνονται ε, λιγότεροι πόροι αλλά για περισσότερα προγράμματα. Οπότε τα σχετικά με τους ε, μη προνομιούχους ε, θα πρέπει να διακρίνεται από κάποιες πιο ανοιχτές, πιο ευέλικτες δράσεις. Και αυτά πρέπει να προσέξουν οι περιφέρειες. Επιζητείται από το κείμενο περισσότερη σύνδεση του σχεδίου και της πρώτας κανονισμού με τον στόχο της οικονομικής συνοχής και της ε, δαφικής συνοχής και της κοινωνικής ούτως ώστε το Ταμείο να μην είναι μέσω τομιακής πολιτικής να συνεχίσει το ΕΚΤ να είναι κάτι το βασικό ως μέσο για την άσκηση της πολιτικής συνοχής και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και το ποιος πρέπει να είναι ο ε, για τις μη προνομικές περιφέρειες και τις, ε, ε τις την απότερη περιφέρεια, όπως λέει το άρθρο εκεί που είναι μειονεκτούσες περιοχές για διάφορους λόγους, για τις περιοχές, ορεινές, ε, ε, μεθοριακές, περαμεθόριες που λέμε. Οπότε θα πρέπει τώρα να δούμε το ότι δεν προβάλλονται αρκετά, δεν προβάλλονται ο ρόλος των περιφερειακών αρχών σύμφωνα με τον κανονισμό. Θεωρείται ότι θα πρέπει να αναδειχθεί το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αρχές για τη διαχείριση του κοινωνικού ταμείου. Μα έχουν την απαραίτητη μεγάλη εμπειρία και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει σχέση με τις δομές της ε, διαχείρισης του ταμείου. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στην διοικητική δομή κάθε κράτους ε, μέλους και ιδίω εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη αποκέντρωση και επίσης ε, συνδέεται με τον κοινωνικό πυλώνα το ταμείο και έτσι να μπορούμε να καλύψουμε κάποιες ε, κοινωνίες με λιγότερες ανισότητες, περισσότερη ισότητα, να επενδύσουμε στον άνθρωπο. Και ιδίω αυτό για εκεί που έχει χτυπήσει περισσότερο η κρίση και πιστεύουμε ότι έτσι ο κόσμος θα αγκαλιάσει περισσότερο το ευρωπαϊκό όραμα. Ε, γι' αυτό σας λέω ότι ε, θα πρέπει να προσεχθούν οι, μη προνομιούχοι, ε, τα άτομα με αναπηρία, οι ανήλικοι, οι νέοι. Χρειάζεται επαρκής πρεχοδότηση και να υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης της απασχόλησης των νέων εγγυήσεις, να καλυφθούν αυτά από το Ταμείο και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τα στατιστικά ε, σε κλίμακα τοπική και περιφερειακή ούτως ώστε να είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι για τις ανισότητες ε, μεταξύ περιφερειών της ίδιας χώρας. Το Ταμείο επίση κάνει ένα άνοιγμα όσον αφορά την καινοτομία της κοινωνίας και αυτό υποσχέται πολλά γιατί θα διέπει την κοινωνική μας πολιτική. Το σχέδιο κειμένου επίσης λέει σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας μας το ότι θα πρέπει αυτό το ταμείο να βοηθήσει για την επιτυχία της βιώσιμης ανάπτυξης. Άμεσα να γίνει η προσπάθεια αυτή, άμεσα να βοηθήσει, γιατί πρόκειται για στόχους που μας καίνε όλους, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως προαναφέραμε, άπαξ και ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή για τη γνωμοδότηση, θέλαμε το κείμενό μας να θεωρεί ότι στο επίκεντρο της προσπάθειας του Ταμείου να είναι ο άνθρωπος, η υγεία, οι νέοι, όλοι όσοι έχουν ανάγκη, οι μετανάστες και επίσης να προασπίζεται τα συμφέροντα των τοπικών περιφερειακών αρχών, να έχουμε σημαντικό ρόλο όσον αφορά την άσκηση πολιτικής του Ταμείου στην κοινωνία μας, στις περιφερειές μας λάβαμε υπόψη ότι πρότεινε κάθε πολιτική ομάδα. Προσπαθήσαμε επίσης να καλύψουμε κάθε πτυχή της πραγματικότητας γιατί θέλαμε αυτή η γνωμοδότηση που είναι τόσο σημαντική για τις ε, ε, περιφέρειες να εγκριθεί σε αυτήν την ολομέλειά μας με όσο γίνεται περισσότερη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος θέλει το λόγο για την γενική συζήτηση. Ουδής ζητεί το λόγο, αλλά ακριβώ έγινε αυτή η συζήτηση προηγουμένω Για να δούμε τώρα τι τροπολογίε που αυτή τη φορά είναι αρκετέ και τα πράγματα είναι τώρα πιο περιπλοκά από ό,τι προηγουμένω. Ένα και δύο μαζί. Δεν υπάρχει ένσταση να το κάνουμε από κοινού υπέρ κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 3. Είναι τεχνικό το θέμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προτείνω να ψηφίσουμε από κοινού τις τροπολογίες 5 και 30. Αν υπάρχει αντίρρηση υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Και τώρα έχουμε την τροπολογία 6. Υπέρ. Ζητεί το λόγο κάποιο κύριο. Ναι, ναι. Το 5. Το 5 απερίφθη. Έτσι δεν είναι. Ναι. 6-6 για το 6. Υπέρ. Κατά. Έγκρινεται 7. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 8. Ε, υπέρ κατά εγκρίνεται Τώρα, από κοινού θα ψηφίσουμε τις εξής τροπολογίες. 9 του εισηγητού και 31 της εισηγητρίας μάλλον. Δεν υπάρχει αντίρρηση υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Οπότε το 9, το 31, 32, 33 και 34 καταπίπτουν. Οπότε πάμε στο 10. Άρα καταπίπτει το 15 μάλλον αν εγκριθεί. Πιέζουν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11. Και καταπίπτει το 12. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Οπότε θα ψηφίσουμε το 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το 13 και το 14 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 15 ήδη έχει καταπέσει και πάμε στο 16 υπέρ κατά απορρίπτεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 19 υπέρ κατά απορρίπτεται κάνουμε επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα τη Απορρίπτεται αυτή η τροπολογία και πάμε στο 20 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 21 υπέρ. Κατά. Παλήθευση ηλεκτρονική. Le vote est clos. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Από κοινού 22 και 23. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Πάμε στο 24 της εισηγήτριας και καταβλήθηκε το 25, 26, 27 και αυτά. Ε, πήγαινε υπέρ του 24. Κατά. Εγκρίνεται από κοινού το 28 και το 29 υπέρ κατά εγκρίνονται έχουν καταπέσει οι επόμενες και πάμε στο 35 υπέρ Κατά. Α, απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Le vote est clos et l'amendement est rejeté. Απορρίπτεται. Η 37. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39 και καταπίπτει 40. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43. Και πιάνεται. Θέλετε να μιλήσετε. Α, για το 43. Ο κύριος Απλώς να σας επισημάνω το εξή. Για αυτούς τους κοινωνικούς δείκτες ή κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη πέραν των άλλων οικονομικών ε, κριτηρίων που θα λεφθούν υπόψη στο μέλλον. Αυτά σημαντικά. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Όταν δηλαδή μιλούμε για αυτήν την ένταξη των μεταναστών, δεν θα πρέπει μόνο να βλέπουμε τη διαφορά, ποιοι πόσοι μπαίνουν, πόσοι βγαίνουν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ένταξη σημαίνει υγεία, στέγαση, παιδεία. Άρα είναι σημαντικό οι παραμεθόριες περιφέρειες να προοικοδοτούνται περισσότερο. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Επομένως, ψηφίζουμε για το 43 υπέρ, κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Le vote est clos et l'amendement... Πέρας. Εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά εγκρίνεται 45 της εισηγήτριας καταπίπτουν οι δύο επόμενες υπέρ κατά εγκρίνεται 47 υπέρ κατά εγκρίνεται 48 υπέρ κατά απορρίπτεται 49 υπέρ κατά εγκρίνεται 50 και καταπίπτει η αρχική 50 αυτή είναι τη σύγκριση υπέρ κατά εγκρίνεται 51 καταπίπτει την επόμενη υπέρ κατά απορρίπτεται 52 υπέρ κατά εγκρίνεται και τέλος η 54 υπέρ κατά εγκρίνεται ψηφίσουμε το σύνολο της γνωμοδότησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομοφόνος και συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην σύνταξη της μην τη διατάξη τώρα έτοιμο πρόβλημα. το επόμενο. Η επόμενη γνωμοδότηση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο τη Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ταμείο Συνοχή. Μίχελ Ράισμπερμαν που είναι ο συγκεκριτή, παρακαλώ να έρθει εδώ πέρα στο Προεδρείο, τόσο ώστε να παρουσιάσει έκθεση. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Έχετε το λόγο, κύριε Σεγητά μου. Dank u wel, voorzitter. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αρχίσω με ευχαριστίες προς όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτή τη σημαντική δουλειά μας για τη γνωμοδότηση. Ήταν πολύ καλή συνεργασία με τους ε, υπαλλήλους και θέλω να ευχαριστήσω τους Γουστάβο Λόπες και την ε, Λούσια Μπέρθερα, τον δικό μου εμπειρογνώμονα, εδώ την παρακαθήμενη κυρία και όλους όσοι συνεισέφερα για τη συγκεκριμένη νομοδότηση. Βλέπετε πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του κειμένου και ευχαριστώ την εμπειρογνώμονα. Κάναμε πολύ καλή συνεργασία επίσης με τους διαφόρους ενεχομένους και εμπλεκομένους και με τους υπαλλήλου και τα μέλη φυσικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και με τους συγητές και τους συνεισηγητές των διαφόρων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί έχουν προχωρήσει πολλοί συζητήσεις εκεί ε, στο συγκεκριμένο τομέα. Και αν δεν το είχαμε εγκρίνει σήμερα το δικό μας κείμενο θα ήταν πολύ αργά. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, και μεγάλη σύμπτωση ε, στη δική μας πρόταση με την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε είναι πολύ καλό να βλέπουμε ότι έχουμε μια τέτοια εταιρική σχέση την οποία εκτιμούμε ε, και έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα, τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες αξίες που προωθούμε και υπερασπιζόμαστε. Ε, ε, τα είπαμε, παρουσία της κυρίας Κρέτσου, τα σημαντικότερα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όλοι έχουμε μια δύσκολη και μακρά ημέρα σήμερα. Ε, διαπιστώνουμε ότι με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, γίνεται ένα μεγάλο βήμα προόδου σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής και την απλούσευση της εκτέλεσής της. Το είπα και προηγουμένως, ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη για όλους. Επίσης, ε, η πολιτική συνοχή αφορά την καθημερινότητα την ίδια των πολιτών μας. Το έχει καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δύο μία που μας απασχολούν βρίσκονται στην ίδια τη βάση στις ρίζες στην κοινωνία. Ας πούμε το Horizon 2020 ή αυτό που θα ονομαστεί στη συνέχεια επενδύστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, InvestEU. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας ε, ακριβώς θα πρέπει να είναι αποδέκτες της πολιτικής την οποία εμείς σήμερα συζητούμε. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες και στην Επιτροπή Κοτέρ και ε, προσπάθησα με τις τροπολογίες του εισηγητή να τις ε, ε, ενώσω, να τις συγκεράσω. Δεν ήταν εύκολο γιατί ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους οι διάφορες τροπολογίες. Ο κύριος Σότιγκερ, ο Επίτροπος, είπε όταν δέχεσαι τις ίδιες φοδρές επιθέσεις από διάφορες κατευθύνσεις, τότε μάλλον καλά τα έχεις πάει και δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. θέλω να σε εξηγήσω μερικά πράγματα τώρα η σημαντικότερη συζήτηση για τις τροπολογίες έχει να κάνει με το ρόλο των περιφερειών στην θεματική συγκέντρωση. Στη γνωμοδότησή μου προτείνω η θεματική αυτή συγκέντρωση ε, να ενισχυθεί περισσότερο και το είπα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει σε επίπεδο πυρεφοριών. Σε επίπεδο περιφερειών αυτό σε κάποια συζήτηση. Αλλά εάν εμείς δεν αναλάβουμε ε, να λύσουμε τα προβλήματά μας στην περιφέρεια, ποιος θα το κάνει. Μετά γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για ποσοστά. Ε, ποιο ποσοστό θα πρέπει να αφιερώνεται στις διάφορες θεματικές ενότητες. Νομίζω ότι καταλήξαμε στον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό ανάμεσα στις διάφορες απόψεις στην Επιτροπή Κοτέρ. Επίσης, υπάρχει και μια σειρά τροπολογιών για το ρόλο κάποιων ευάλωτων περιφερειών, των άκρως απομακρυσμένων και άλλων ε, με διάφορες εξαιρέσεις που θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να γίνονται. Είναι κατανοητό γιατί το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολλές περιπτώσεις ζητάει κάτι ειδικό, αλλά δεν εξηγεί τι εννοεί. Αυτό το θεωρεί πλεονέκτημα γιατί όταν κάτι είναι ασαφώς διατυπωμένο χωράει και πολλές ερμηνείες και προσαρμογές, ο καθένας στα μέτρα του. Και όταν ο ευρύ ε, ορισμό η ευρεία περιγραφή αντικαθίσταται από ένα μακροσκελή κατάλογο με ειδικέ εξαιρέσει, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και περιπλέκονται. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να μην ε, ε, δυσκολέψουμε το κείμενο άσκοπα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία να τα λέμε με το όνομά τους και να μας βοηθούν για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Αλλιώ θα αποδυναμωθεί η γνωμοδότηση. Αυτά, Πρόεδρε, και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί το λόγο για τη γενική συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση αυτήν όχι μόνο είναι σημαντική χρηματοδότηση για τις περιφέρειες, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τις ε, νέες ευκαιρίες απασχόλησης που πρέπει να δημιουργηθούν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέλη της Επιτροπής μας δείχνουν μέσω της γνωμοδότησης αυτής πώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει πόλεις, περιφέρειες σε πάρα πολλούς τομείς. Θα πρέπει να καταφέρνουμε να προβάλλουμε περισσότερο τα θετικά αποτελέσματα, τα διαρθρωτικά ταμεία, θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν ως τελικό παραλήπτη τις περιφέρειες και θα πρέπει να στείλουμε χειρό μήνυμα προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τα κράτη-μέλη. Με την συμμαχία αυτή για την πολιτική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών κατάφερε πραγματικά να δείξει πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα διορθωτικά ταμεία και το θετικό αντίκτυπο που έχουν επιτόψει. Ευχαριστώ πολύ και υποστηρίζω αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία των τροπολογιών. Η τροπολογία παρελθόν 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 του εισηγητή και καταπίπτουν οι αρχικές 4 και 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 του εισηγητή που και καταπίπτουν οι 6 έως 8 υπέρ κατά ε, εγκρίνονται. Η τροπολογία 9 του εισηγητή καταπίπτουν οι 9 έως 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 13 του εισηγητή καταπίπτουν 13 και 14 υπέρ κατά Όχι συγκρίνονται. Η τροπολογία 15 του εισηγητή καταπίπτουν οι 15, 16, 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η τροπολογία 19 του εισηγητή και αν εγκριθεί καταπίπτουν οι 19 και 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 20, συγγνώμη, υπέρ κατά απορρίπτεται. Η τροπολογία 21 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η τροπολογία 22 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η τροπολογία 23 υπέρ κατά απορρίπτεται 24 υπέρ κατά απορρίπτεται το σύνολο τώρα της γνωμοδότησης υπέρ τελική ψηφοφορία κατά αποχές εγκρίνεται η γνωμοδότηση επίσης ομόφωνα συγχαρητήρια κύριε Σιγητά Le prochain avis Περνάμε στην επόμενη γνωμοδότηση που έχει να κάνει με την πρόταση κανονισμού που δημιουργεί ειδικέ ε, διατάξεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Πρόκειται για το πρόγραμμα που είναι γνωστό με το όνομα Interreg. Να καλέσω την συντάκτηρα της γνωμοδότης, την συγγήτριά μας, μάλλον την Μαρία Αντουανέτ Μομπερτιούς, θα της δώσω ευθύς αμέσως το λόγο μόλις φτάσει εδώ στο Προεδρείο. Ναι. Merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, που είναι γνωστή με το όνομα Interreg, είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα πολιτικά εργαλεία για τους πολίτες. Μας επιτρέπει να έχουμε ανταλλαγή εμπεριών και δράσεων μεταξύ τοπικού και περιφερειακού επίπεδου και κεντρικού επίπεδου για μία η Ήπειρο η οποία έχει τα περισσότερα ιστορικά σύνορα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία αυτή προκειμένου να έχουμε οικονομική, δαφική, κοινωνική συνοχή μεταξύ των περιφερειών μας, αλλά για να καταφέρουμε να συνεργαστούμε και με τις παραμεθόριες τρίτες χώρες πέρα από τα εξωτερικά μας σύνορα δηλαδή. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα αυτό. Το είδα αυτό τους τρει τελευταίου τελευταίους μήνες και κατά τη διάρκεια όλων των Συζητήσουν και συναντήσεων που είχαμε επιτόπου. Σήμερα λοιπόν μιλάμε όχι μόνο για τους τεχνικούς κανονισμούς και ρυθμίσεις, αλλά για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη, γενικότερα για ένα όραμα μιας Ευρω... Ενωμένης Ευρώπης, η οποία στο πλαίσιο ότι θα έχει σχέδια επικοδομητικής συνεργασίας, που θα επιτρέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προσπάθησε να απλουστεύσει περισσότερο τους κανονισμούς και να προωθήσει τη συνέργεια, ιδίως με τις τρίτες χώρες. Περιλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο άρθρο όσον αφορά τα μικρά έργα, πρωτοβουλία που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή των Περιφερειών, μικρά έργα που ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αναγνωρίζονται οι συγκεκριμένε ιδιαιτερότητε των εξόχω απόκεντρων περιφερειών μέσω μια νέα συνιστόσα 3, που ουσιαστικά εδώ πέρα για πρώτη φορά καταφέρνουμε να καλύψουμε τον άγκη αυτή. Προβλέπεται ότι μπορούμε να έχουμε διαπεριφερειακές επενδύσεις και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο τις δράσεις των περιφερειών εκείνων που έχουν επενδύσει περισσότερο στις ευφύς επενδύσεις και τεχνολογίες όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος Μάρκο Μάρκολα πριν από λίγο. Στα πλαίσια της Επιτροπής Κοτέρ επίσης, είδαμε ότι ορισμένα σημεία του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να βελτιωθούν ε, αν πραγματικά θέλουμε η ευρωπαϊκή αυτή εδαφική συνεργασία να είναι υποφελή για όλες τις περιφέρειες, αν θέλουμε να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και αν θέλουμε τελικά να απορρέει από μια λογική πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και αν θέλουμε να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Όπως είπε η Επίτροπος ε, Κρέτσου πριν από λίγο, θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε μια Ευρώπη πιο κοντά στου πολίτε η πρωτοβουλία και η πρόταση, αν θέλετε, το ρώσιμο που προωθούμε μέσω τη γνωμοδότηση αυτή στην Επιτροπή Κοτέραντα και σήμερα και με συνεργασία με τον βουλευτή Αγιμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόταση η οποία εγκρίθηκε μάλιστα και στην Επιτροπή Ρέτζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά και σε σχέση με την έκθεση Μαρίνη Σνάιντερ που εγκρίθηκε πριν από λίγο. Η πρώτη λοιπόν αυτή πρόταση είναι ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Συνεργασία θα πρέπει να περάσει από τα 50% στο 3% του συνολικού προπολογισμού της πολιτικής συνοχής και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την πολιτική της παραδοσιακής συνεργασίας και ιδίω στο πλαίσιο του Interreg Ευρώπη που αντιστοιχεί μόνο στο 0,1% του συνολικού φακέλου της πολιτικής συνοχής. Δεύτερη πρόταση θέλουμε το επίπεδο σε χρηματοδότηση να περάσει από το 70% στο 85%. Υπάρχουν πολλοί παράγοντε επιτόπου που μα το απέτησαν αυτό, μα το ζήτησαν. Θέλουμε επίση ένα επιπλέον προπολογισμό 0,3% από τη συνολική χρηματοδότηση πολιτική συνοχή. σε συμφωνία με τον Ευρωβουλευτή Αριμό αλλά και με τους εισηγητές Μαρίνη Σνάιντερ το αποφάσισαμε αυτό για να συγχρηματοδοτήσουμε ένα νέο εργαλείο διαπεριφερειακής συνεργασίας για την καινοτομία αυτή τη φορά ένα δισεκατομμύριο ευρώ θέλουμε να έχουμε για την καινοτομία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε επίσης να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για αυτό το εργαλείο. Αυτό προτείνουμε στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ακριβώς επειδή υπάρχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για το εργαλείο αυτό και ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι διαφέρει από την παραδοσιακή ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προτείναμε μια συμβαστική τροπολογία με τη συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων εγκρίθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες αυτή η τροπολογία και θα την παρουσιάσουμε σε λίγο. Προβλέπει ότι το νέο αυτό εργαλείο, το νέο αυτό μέσο θα πρέπει να είναι ανοιχτό προ όλε τι περιφέρειε Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ή τις περιφέρειες εκείνες που αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς ή διαρθρωτικού περιορισμού. Τώρα, όσον αφορά την θαλάσσια συνεργασία, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας. Το είπα πάρα πολλές φορές αυτό. Ένα σύνορο, ότι είναι χερσαίο ή θαλάσσιο, με σύριγγα ή γέφυρα ή άνευ, παραμένει ένα σύνορο. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν και θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Στο πλαίσιο επίση του Brexit, ζητήσαμε η πολυεπίπεδη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρηθεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας σύνδεσης όπως αυτή που έχουμε με την Νορβηγία. Προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις των Βρετανών φίλων μας. Εν κατακλείδη, αποδεχθήκαμε όλες τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες συνάδουν με τις προτάσεις αυτές, υπερψηφίστηκαν στην Επιτροπή Κοτέρ, με την πλειοψηφία των περισσότερων πολιτικών ομάδων καταλήξαμε σε κάποιες συμβαστικέ προτάσεις τι οποίες θα πρέπει τώρα να ψηφίσουμε. Θα ήθελα ολόθερμα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες που συνέβαλαν στην εμπλουτιστή πρόταση αυτή, να ευχαριστήσω το προσωπικό της Επιτροπής ΚΟΤΕΡ, να ευχαριστήσω επίση του εμπειρογνώμονε μα, οι οποίοι άκνα, άοκνα με συμμετείχαν στην εκπόνηση της γνωμοδότησης αυτής και να ευχαριστήσω επίσης όλους τους τοπικούς και περιφερειακούς ηθήνοντες οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπόνηση της γνωμοδότησης αυτής καθότι ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και οι οποίοι με την καθημερινή τους εργασία συμβάλλουν πάρα πολύ στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Μακάρθη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την η συγκίτριά μα για την εκπόνηση του σχεδίου αυτού γνωμοδότησης. Το πρόγραμμα Interreg είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις περιφέρειες Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία δύο χρόνια στη δική μου την περιφέρεια είδαμε ότι είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα μέσω τη Ευρωπαϊκή αυτής εδαφική Συνεργασία με άλλε δηλαδή περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καταπληκτικό το πρόγραμμα Ίντερεκ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιοδήποτε δήμαρχος, ευρωβουλευτή, βουλευτής ή απλό πολίτη θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Το πρόγραμμα Ίντερεκ έρχεται και λύνει τα πιο πολύπλοκα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι περιφέρειε Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί πραγματική ελπίδα όσον αφορά την μελλοντική ανάπτυξη των περιφερειών μας. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Μάικλ Γιούγκου Αγκεζάγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πρώτα που να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Κατά 95% συμφωνούμε. Το ξέρει. Έχουμε όμως σε συγκεκριμένο θέμα διαφωνία όσον αφορά το συντελεστή 5 είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διαπεριφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη και πολλές περιφέρειες έχουμε σχετική εμπειρία στο πλαίσιο των θεματικών πλατφορμών. Ε, θα ήθελα να προσέξουμε το εξή. Μας είπατε ότι έχουμε ε, κάποιους συμβασμούς τελευταίες Είπατε να ψηφίσουμε από κοινού το, το 10 ρο και το 18 ρο. Αυτό είναι καινούριο φρούτο, γιατί όπως είπατε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα σε επιτροπή ενέκρινε τη συμβαστική διάταξη όσον αφορά την πρόταση εδαφικής συνεργασίας. Εκεί, σε αυτή τη συμβαστική διάταξη του Κοινοβουλίου, αυξάνει το Κοινοβούλιο την πρικοδότηση για το ΡΕΓ. 10% ε, περισσότερο από όσο προβλέπει η έκθεση. Και έχουμε τώρα το παράδοξο η Επιτροπή των Περιφερειών να ζητεί λιγότερα χρήματα από ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα όπως το Ίντερνετ Γι' αυτό λέω, αναθεωρήστε σε σχέση με την ψηφορία για το 10 και το 18 ρο. Εγώ θα καταψηφίσω. Μας τα είπατε η συγκεντρία. Ίσως να μην εγκριθούν αυτές οι διατάξεις, αλλά θα πρέπει να αυθυγραμμιστούμε με αυτό που ζήτησε πριν από δύο μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό σας λέω να αναθεωρήσετε και να καταψηφίσουμε αυτές τις δύο ε, τροπολογίες, με τις οποίες διαφωνώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Και τώρα. Ζανέτ Μαγιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σημαντικό θέμα. Σημαντική και η έκθεση. Έχουμε πει πάρα πολλά όσον αφορά αυτό το συντελεστή, το στοιχείο 5, όσον αφορά τι ε, επενδύσεις για την καινοτομία, για το Interreg. Και έχουμε το 18ο τη εισηγήτρια ω ε, τροπολογία. Προσοχή. Μην χάσουμε αυτό το μέσο ούτω ώστε να υπάρξει συνεργασία σε όλε τι περιφέρειες. Ναι, καλύπτει όλε τι περιφέρειες μην χαθεί αυτό το μέσο που αφορά τον εξυγχρονισμό στη βιομηχανία που το χρειάζεται η Ευρώπη. Και όπως είπαμε στις 3 Δεκάτου η Περιφερειακή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε για υυξημένη προϋποδότηση. Γιατί εμείς να μην το κάνουμε το ίδιο. Άρα εμείς να εγκρίνουμε το 18 και να καταψηφίσουμε τα 15 και 18. Λουκ Φαντεμπράντερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω τους δύο συναδέλφους και τα επιχειρήματά τους. Θέλω όμως να πω ρητά και στο εξής. Σας παραπέμπω σε μια πρωτοβουλία που συμμετέχουν ε, και βελγικές περιφέρειες και σύνολο 43 ενότητες για μια ε, διασυνοριακή συνεργασία με κοινοτομία. Όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να δούμε ε, να συμμετέχουν εκεί όχι μόνο οι διοικητικέ περιφέρειες, αλλά και περιφέρειες που σε λειτουργικό επίπεδο ε, είναι συναφείς. Υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα. Ας πούμε, Λέβεν, ε, Έιτχόβεν, Άχεν. Είναι ένα τρίγωνο καινοτομία και θα ήταν πραγματικά μοιραίο σφάλμα αν δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε στην πέμπτη ε, Συνιστώσα, παρόλο που δεν είμαστε διοικητικά ε, συνδεδεμένες περιφέρειες. Είναι σημαντικό να επανέλθει η συνιστόσα 5. Αλλιώς, πραγματικά θα έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες και θα χάσουμε μεγάλες ευκαιρίες. Να το κοιτάξει παρακαλώ η συγγήτρια ξανά και να το συμπεριλάβει στην γνωμοδότησή της. Σας ευχαριστώ. Je ne vois pas d'autres demandes de parole, alors je... Δεν ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Θα ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγητρία μας, παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχάς να σε επενθυμίσω ότι εδώ πέρα διακυβεύονται πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία στον θαλάσσιο τομέα όσον αφορά την διατήρηση της συνιστώσας 3 που αφορά πάρα πολλές περιφέρειες που υπάγονται στο πρόγραμμα Interreg, θα έλεγα όλες τις περιφέρειες, και έπειτα έχουμε και τη συνιστόσα 5 που είναι εξίσου σημαντική. Για τα τρία αυτά σημεία διεξήχθηκαν σημαντικότατες συζητήσεις στην Επιτροπή Κοτέρα και μετά τις συζητήσεις αυτές, μετά από αίτημα των εκπροσώπων, των εμπλεκόμενων περιφερειών στο σχέδιο Vanguard, αποφασίσαμε να καταλήξουμε σε μία συμβαστική πρόταση η οποία εκπονήθηκε βάσει της εξής λογικής. Από τη μία πλευρά να έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για τη διαπεριφερειακή καινοτομία, και εμείς προφανώς εμείς υποστηρίζουμε τη συνιστόσα 5, απλώς στη σφαιρική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ζητάμε μέσω της συμβαστικής αυτής τροπολογίας να έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο θα στοχεύει ακριβώς τη νέα αυτή μορφή συνεργασίας που δεν είναι παραδοσιακή μορφή συνεργασίας. Έχουμε μια πρωτοβουλία συγκεκριμένη, στοχευμένη, υπέρ της καινοτομία. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται εκεί είναι εντελώ διαφορετικοί από αυτούς που χρησιμοποιούν παραδοσιακά για τη διαπεριφερειακή συνεργασία στα πλαίσια των Interreg. Επίσης, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επισημοποιήσουμε, όπως ακριβώς έγινε με στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως ακριβώς έγινε και στο πλαίσιο της έκθεσης Σνάιντερ Μαρίνη, μπορούμε να επισημοποιήσουμε και να παγιώσουμε ένα ποσό ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να το επαναλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν κινδυνεύει καθόλου η συνιστόσα 5. Αν το αντίθετο μάλιστα, έχουμε πλέον για τη συνιστόσα αυτή ειδικό κεφάλαιο με ειδική χρηματοδότηση και την Παρασκευή το απόγευμα το Συμβούλιο έκρινε και αυτό ότι η συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί βάσει των, του, Ταμείου, Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση που έγινε από τον ΚαΕΛΑ, στην ίδια πολιτική ομάδα ανήκουμε, το τελικό ποσό είναι πάνω κάτω το ίδιο. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εμείς κάτω από αυτό το οποίο έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως σας είπα, εργαζόμαστε πάρα πολύ με τον Ευρωβουλευτή κύριο Αγιμό, επομένως έχουμε συντονιστεί και στο ζήτημα του ποσού και προτείνουμε 10 δισεκατομμύρια για την παραδοσιακή διαπεριφερειακή συνεργασία όπου θα περιλαμβάνονται εκεί πέρα όλες οι συνιστώσεις οι παρελθούσες και θα έχουμε έπειτα και αυτό το 1 δισεκατομμύριο, 900 περίπου εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά το νέο αυτό που θα έχει να κάνει με την καινοτομία. Τέλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάχθηκε τελικά με τη δική μα την άποψη, γιατί Δευτέρα το απόγευμα στην Επιτροπή Ρέτζι αποφάσισε ότι θα πρέπει να ενσωματώσει το σύνολο των περιφερειών, ακόμα και τι λιγότερο αναπτυγμένε για την πρωτοβουλία αυτή. Η καινοτομία δεν μπορεί να αφορά συγκεκριμένε μόνο και λίγε περιφέρειες στην Ευρώπη. Η καινοτομία είναι τεχνολογική, αλλά είναι και κοινωνική και θα πρέπει να επιτρέπει σε όλες τι περιφέρειες να μπορούν να συγκλίνουν προ ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξη. Αυτά είχα να σας πω λοιπόν υπέρ των τροπολογιών, υπέρ της τροπολογίας 25. Όσον αφορά τώρα την 10 και 18 άρα, αποτελούν απόρριο ουσιαστικά των τροπολογιών που κατέθεσε ο Μικαέλα. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε τώρα στις τροπολογίες, λέει ο Πρόεδρο. Σας προτείνω από κοινού τις 1-4 να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 5 άρα αντικαθιστά την αρχική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 άρα καταπίπτει την, ε, κάνει να καταπέσει 6 και 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 και 9 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται. Προτείνω να ψηφίσουμε από κοινού την 10R και 18 άρα, γιατί έχουν σημαντικές συνέπειες. Θα καταπέσουν οι 10, 11, 12, 13, 24, 45, 46, 18, 19 και 20. Όλες αυτές καταπίπτουν εφόσον εγκριθούν οι 10 και οι 18 άρι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Περνάμε έτσι στην τροπολογία 15 άρα καταπίπτουν 15 και 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. Περνάμε έτσι στην τροπολογία 21 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 22 και έτσι καταπίπτει 23 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 λοιπόν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 25 όπου έχουμε μία προφορική συμβαστική τροπολογία η οποία εγκριθεί οι 26, 27 και 28 καταπίπτουνε να ζητήσω από την εισηγήτρια να μας εξηγήσει την προφορική συμβαστική τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, στην, στις τελευταίες αυτές τροπολογίες ήρθαν σε επαφή μαζί μου εκπρόσωποι από τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες που δεν είχαν συμμετάσχει στην Επιτροπή Κοτέρ και θέλανε από νομικής πλευράς να μπορούν να καλυφθούν από την τροπολογία αυτή. Θέλανε να γίνει ρητή αναφορά στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες. Ήρθα σε επαφή με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, συμφώνησαν μαζί μου και κατά αυτόν τον τρόπο υποβάλαμε την τροπολογία αυτή που ουσιαστικά έχει να κάνει με τη γλωσσική διατύπωση. Υπέρ με τη συμβαστική τροπολογία, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τη τροπολογία 29, καταπίπτουν οι 30 και 31 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30, λοιπόν, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 30. Άρχη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32, γιατί κατέπεσε 31, υπέρ 32 παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 και έτσι καταπίπτει 34 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35 και έτσι καταπίπτει η 36, 37 και 51 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 36 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 37 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 38 υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία 39 και έτσι καταπίπτει 40 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε έτσι στην τροπολογία 47, Απέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48 και 49 είναι ταυτόσιμες. Τις ψηφίζουμε μαζί λοιπόν υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση και τροπολογία 52 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία. 53 και 54 μαζί, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία υπέρ της γνωμοδότησης παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και σε όλους τους συνεργάτε της. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο 9. Μικρό αδερφάκι του 8 ουσιαστικά ε, είναι γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού σύμφωνα με τη δημιουργία ενός διασυνοριακού μηχανισμού. Ε, Η συγγετής είναι ο συνάδελφός μας ε, Μπάουκε Άρεντς και τον καλό να έρθει στο Προεδρείο. Monsieur Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μου και ε, ιδιαίτερα τη Γραμματεία της Επιτροπής ΚΟΤΕΡ για την υποστήριξη και τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Πάρα πολλή δουλειά έχουν κάνει και με έχουν υποστηρίξει τα μάλα. Πολύ ε, επικοδομητική συνεργασία είχα και με τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Εγώ είμαι δημοτικό σύμβουλο σε μια παραμεθόρια περιοχή στα σύνορα Ολλανδίας και Γερμανία. και πραγματικά πρέπει να σα πω ότι οι περιοχέ αυτέ ανθούν και έχουν μεγάλο δυναμικό. Τα τελευταία χρόνια με την χρηματοδότηση ε, του Ιντερεκ ε, είχαμε πολλά έργα από κοινού ε, με επιτυχία και αντιμετωπίσαμε πολλές καταστάσεις. Αλλά το σύνορο σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει εμπόδιο ε, για ομαλή συνεργασία και γρήγορη. Κυρίως υπάρχουν διοικητικά και νομικά εμπόδια. Ε, χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για να τα λύνει αυτά. 30% ε, των κατοίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σε παραμεθόριες περιοχές, εργάζονται, πηγαίνουν σχολείο, κάνουν ψώνια και τους εμποδίζουν αυτά τα σύνορα, τα εμπόδια ή διπλές ε, διαδικασίες ή περίπλοκες διαδικασίες. Γι' αυτό με τη συγκεκριμένη πρόταση θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, να πέσουν αυτά τα εμπόδια και οι φραγμοί διοικητικοί και οι νομικοί. Και κυρίως είναι εθελοντικός μηχανισμός. Από τις ε, περιφέρειες μπορούμε να βρούμε κοινέ λύσεις για ένα ειδικό έργο κάθε φορά. Αλλά θα πρέπει να ψάχνουμε τι νομοθεσία ισχύει στη γειτονική χώρα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου το 2015 του Συμβουλίου που εμπνεύστηκε αυτή την πρωτοβουλία για ένα κανονισμό ε, που δίνει τη συνοριακή δυνατότητα μάλλον στις περιοχές αυτές να συνεργάζονται καλύτερα. Υπάρχουν ε, εργαλεία, υπάρχουν τροπο, πρωτοβουλίες και μπορεί να δημιουργηθεί και αυτός ο μηχανισμός. Εκεί μπορούμε να βασιστούμε, να πατήσουμε στα καλά παραδείγματα που υπάρχουν, όπως είναι ε, η Ένωση Benelux και το Βόρειο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την Επιτροπή Κοντέρ, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όλα τα αρμόδια όργανα που συνεργάστηκαν προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλω να τονίσω τα εξή σημεία. Ε, μια πιο ξεκάθαρη στρατηγική επικοινωνίας είναι απαραίτητη για να διασκεδάσει φόβους και αμφιβολίες. Ε, θα πρέπει να μπορούμε ε, να προχωρούμε σε ταχεία εφαρμογή των έργων και επίσης να έχουμε καλούς μηχανισμούς για να μπορούν να αξιολογούν κατά πόσο ο κανονισμός λειτουργεί σωστά στην πράξη. Έτσι θα προχωρήσουμε για να έχουμε όσο γίνεται καλύτερες λύσεις. Το Συμβούλιο Υπουργών τώρα και κάποια κράτη-μέλη αμφιβάλλουν και μεταξύ αυτών και η Ολλανδία για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου το υποστηρίζει αυτό ως πρόταση, αλλά και εκεί ακούγονται αμφιβολίες. Πρέπει να βοηθήσουμε τις παραμεθόριες περιοχέ και χρειάζεται επιγόντως και γρήγορα αυτός ο μηχανισμός. Θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε τη σημερινή πρόταση και Θέλω να ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους σχεδόν από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία που είχαμε στην Επιτροπή ε, ΚΟΤΕΡ με επικοδομητική συνεργασία. Και ευχαριστούμε και για τις τροπολογίες. Ε, υπάρχει ευρεία υποστήριξη της Επιτροπής ΚΟΤΕΡ για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο θέλει το λόγο, ευχαριστώ πολύ στη γενική συζήτηση τώρα. Ουδή ε, από ό,τι βλέπω. Α ψηφίσουμε λοιπόν τι τροπολογίε. Η τροπολογία υπαριθμών 1. Μαζί με τις τροπολογίες 3, 9 και 10. Και αν εγκριθούν όλες αυτές, καταπίπτουν οι τροπολογίες 2 και 13. Ψήφι υπέρ παρακαλώ κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 4. Προτείνεται με αλφαγιώτα να ψηφιστεί μαζί με την 6 και τη 12. Ψήφι π. Κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά εγκρίνεται η 15 υπέρ κατά εγκρίνεται η τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αυτή υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται ομόφωνα γνωμοδότηση και συγχαρητήρια στον εισηγητή και ας ελπίσουμε η έκκληση που απευθύνει στις κυβερνήσεις αυτή η γνωμοδότηση να εισακουστεί. Την υποστηρίζω προσωπικά απολύτως γιατί γνωρίζω πολύ καλά την προϊστορία αυτού του ε, μέσου και του εύχομαι κάθε επιτυχία. Πάμε στο σημείο 10 τώρα της ημερήσιας διάταξης και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα πάνε τόσο ομαλά και τόσο γρήγορα όπως με το 9. Έχουμε τη γνωμοδότηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα καλέσω εδώ τον συνάδελφό μας, εισηγητή κύριο Γκυγιόμ Χος.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 Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, συγγνώμη, υπήρχε ένα πρόβλημα ενημέρωση επικοινωνία. Euh, πρώτα, πρώτα ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν για να συντάξουμε αυτήν την ε, έκθεση. Είναι σημαντική όπως είναι σημαντικές και πολλές άλλες που εδώ διεκπαιρεώνουμε, αλλά αφορά την πρώτη κοινοτική πολιτική, την γεωργική πολιτική. Βεβαίω έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες. Αλλά οι λίγες εκατοντάδες δικές μας βγαίνουν μία μπροστά στο κοινοβούλιο που είχε 7.000 αντίστοιχες. Οπότε υπήρξε αυτή η συμμετοχή, είναι σημαντικό το θέμα, αλλά είναι και το αποτέλεσμα των προσπαθειών με το επιτελείο της Επιτροπής μας και με τον εμπειρογνώμονά μου. Οι βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής μας είναι να έχουμε μια οικογενειακή, βιώσιμη πολιτική παντού για όλες τις ε, περιφέρειες. να καλύψουμε την εδαφική συνοχή σε πόλεις, την Ήπεθρο, οι στόχοι οι οποίοι καλύπτονται από την συνθήκη της Λισαβόνας. Πέρσι εγκρίναμε την μεταρρύθμιση και είπαμε όλοι εδώ να υπάρχει μια ΚΑΠ δίκη βιώσιμη, αντιλέγγυα και να παραμείνει κοινή. Οι τροπολογίες μου ακριβώς αυτό κατατείνουν πιο δίκαιη. Θα πρέπει να πάρει πιο δίκαιη κατανομή όσον αφορά τις ε, ενισχύσεις. Σας υπενθυμίζω, 3% των γεωργών παίρνουν το 50% των ενισχύσεων και το 20% το 80% των ενισχύσουν επομένω, θα πρέπει να γίνει δικαιότερη κατανομή. Και στο κείμενο μιλούμε για εξωτερική εσωτερική σύγκληση, μιλούμε για καινούργια άνω όρια όσον αφορά τις ενισχύσεις, μιλούμε για διανεμητικές καταβολές, πληρωμές, περισσότερο για το πρώτο εκτάριο και να είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα που να χρησιμοποιούνται, υποχρεωτικές ρυθμίσει και επίσης ενίσχυση στις μικρές εκμεταλλεύσεις υποχρεωτική για τα κρατημέλη. Γιατί αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις κρατούν ζωντανή την ύπεθρο ε, και δημιουργούν απασχόληση. Θέλουμε να είναι πιο βιώσιμη ε, σε σχέση με το κλίμα, σε σχέση με το περιβάλλον. Στόχοι σε σχέση με την έκθεση του ΟΗΕ που έλεγε ότι θα πρέπει να μειώσουμε περισσότερο το αέρια θερμοκηπίου και η γεωργία έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό αιτήσια κυκλική εναλλαγή των καλλιεργιών ε, προσαρμοσμένη στην αιρεσιμότητα και να υπάρχει αντιστάθμιση πέραν της αιρεσιμότητας αύξηση σημαντική ε, το και λιγότερα ζυζανιοκτώνα και να έχουμε επίσης οικολογική ε, ενίσχυση και να μην υπάρχει κτηνοτροφία σε κλουβιά. Επίσης χρειαζόμαστε κάποιες δίκαιες σταθερές τιμέ στη Γεωργία. Ακριβώς όπως είπαμε στην τελευταία φορά η ρύθμιση της αγοράς σημαίνει ότι τώρα υπάρχουν ε, πιο μεγάλες ε, δαπάνε. Θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτά που είπαμε σε περίοδο κρίσης και να υπάρχει τώρα ένα μοντέλο πιο ποικίλο και πιο ανθεκτικό. επίση. να ενισχύσουμε την υπέθρο, να υπάρχει ανάπτυξη τη υπέθρο με συγχρηματοδότηση και να μην μειωθούν οι προποδοτήσει και να τι πλαισιώσουμε τι εκμεταλλεύσει και έτσι να υπάρξει η μετάβαση προς βιωσιμότητα με τον δεύτερο πυλώνα και με επενδύσει θα πρέπει προς τα εκεί να κατατείνουμε. Ποιότητα, ε, διατροφή, ορεινή κτηνοτροφία, όλα αυτά να υποστηριχτούν και όλα αυτά είπαμε ότι αφορούν την δημόσια υγεία και την ύπεθρο. Οπότε θα πρέπει να, να αλλάξουμε τα μέσα πολιτικής και έτσι να βρούμε κάποια μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η νέα κάπου να είναι πραγματικά κοινή. Τα στρατηγικά εθνικά ε, προγράμματα θα πρέπει να κατατείνουν στην ε, βοήθεια της περιβαλλοντικής πολιτικής. Και για αυτό έχω κάνει κάποιες τροπολογίες με αριθμητικές προτάσεις για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά να αντιστοιχούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Εάν αυτές οι απαιτητικές κάποιες φορές προτάσεις, ε, αλλά απαραίτητες κατά την άποψή μου, ε, για να διατηρηθεί ο προπολογισμό τη κάρτα που εδώ που θέλουμε. Ε, νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που έχουμε αναλάβει για να υπάρχει μια δίκαιη, ε, βιώσιμη και αλληλέγγυα ΚΑΠ. Γι' αυτό, συνάδελφοι, σας ζητώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου για το κείμενο της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής μας. Μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Γενική συζήτηση τώρα. Έχουν εγγραφεί πρώτος ο κύριος Μπιάνκο. Πρόεδρε, γνωρίζω πολύ καλά έχοντας συμμετάσχει στα πράγματα της Επιτροπής των Περιφέρειων από τότε που ιδρύθηκε ότι η αγροτική πολιτική είναι ένα θέμα για το οποίο η Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και το ίδιο Ευρωκοινοβούλιο και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα έχουν μεγάλες διαφωνίες μεταξύ τους και πολλές φορές η συζήτηση είναι και περίπλοκη. Αναγνωρίζω ότι σήμερα η συζήτηση θα είναι ακόμη πιο δυσχερής διότι η γνωμοδότηση αυτή δεν ε, βρέθηκε στην Επιτροπή της. Ε, επειδή υπάρχει υψηλό αριθμό τροπολογιών, θα έπρεπε να είχε εξεταστεί εντελεχέστερα από την αρμόδια επιτροπή. Τώρα βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική στιγμή. Η Ιταλική αντιπροσωπεία, και το λέω εξ ονόματο ε, τη Ιταλική αντιπροσωπεία, και όχι μόνο εκφράζοντα την προσωπική μου άποψη ω μέλο των σοσιαλιστών. Η Ιταλική αντιπροσωπεία αποφάσισε σήμερα στην τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα να ακολουθήσει τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής των Περιφερειών σε σχέση και με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Είναι πολύ θετική η γνωμοδότηση του εισηγητή για κάποιες πτυχές, αλλά για κάποιες άλλες είναι εντελώς το αντίθετο. Δεν ε, λαμβάνει υπόψη κάποιες απαιτήσει του κόσμου της γεωργίας, της αγροτιάς, και το πώς πρέπει να ε, μεταλλαχθεί ανάλογα με τις σύγχρονες ανάγκες. Το λέω εκ μέρου τη Ιταλική Αντιπροσωπεία, λοιπόν. Η τελική μα ψήφο θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει με τι τροπολογίε. Προτείνω στου συναδέλφου να κοιτάξουν με μεγάλη προσοχή την κάθε μια τροπολογία ξεχωριστά, διότι ορισμένε τροπολογίε του εισηγητή φαίνεται να επηρεάζουν άλλε τροπολογίε που έχουν υποβάλει μεμονωμένα μέλη της Επιτροπής τη ε, Επιτροπή των Περιφερειών. Το ε, επισημαίνω λοιπόν γιατί είναι σημαντικότατη η συγκεκριμένη ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο συνάδελφος Μαρτίνες Αρεγκουή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά οι τροπολογίε δείχνουν τον αριθμό τη πόσε ανησυχίε μα προκαλεί όλη η συζήτηση για την κοινή γεωργική πολιτική. Η πρόκληση είναι να ορίσουμε μια σύγχρονη κάπα πιο ευνόητη, πιο δίκαιη για όλου. Όπω ε, είπε και ο εισηγητή, ε, που θα εγγυάται την ανταγωνιστικότητα του τομέα με τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση των γεωργικών υποδομών, εξονισμό των ε, εκμεταλλεύσεων και το γεωργοδιατροφικό κλάδο. Επίσης, ανάπτυξη ε, του ε, υπαίθρου και καταπολέμηση απερίμωσης. Είναι μεγάλη ανησυχία μας αυτή. Δεν πρέπει λοιπόν να γίνουν περικοπές ή αν γίνουν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ λίγες και τελικά ένα μεγάλο τμήμα ε, των στρατηγικών σχεδίων ε, των ε, κρατών μελών εξαρτάται, έχει να κάνει τη γεωργία, πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τη νεολαία. Αν θέλουμε να ανανεωθεί ηλικιακά ο πληθυσμός των αγροτών, θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς για να αποφύγουμε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται να συνεχίσουν να παίρνουν τις άμεσες ενισχύσεις από την κοινωνική πολιτική γιατί αλλιώς ε, δεν θα μπορέσουν νέοι να ασχοληθούν με τη γη. Οι ενισχύσεις οι οποίες σχετίζονται με σημαντικούς τομείς που έχουν προσθέμενη αξία, όπως είναι ο, είναι ο παραγωγικός ε, τομέας, έχουν μεγάλη παραγωγική αξία. Θα πρέπει να γίνουν ε, σεβαστές ιδιαιτερότητες όταν μιλάμε και για το παραγωγικό δυναμικό. Και πρέπει να βοηθήσουμε, όπως είπα, να καταπολεμηθεί η απερίμωση. Αυτή η περικοπή του 15% ουσιαστικά αφαιρεί, στερεί αξία από αυτές τις πολιτικές που θέλουμε να προωθήσουμε για την καταπολέμηση της αστιφιλίας και πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν νέοι πόροι στα σχετικά γεωργικά ταμεία. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. La parole... Ευχαριστώ πολύ. Jacques Blanc. Je veux Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πολύ σημαντική η εργασία του. Το θέμα είναι πολύ απαραίτητο και σημαντικό για το μέλλον του ευρωπαϊκού μοντέλου χωροταξίας μέσω της διατήρησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ευρωπαϊκή επικράτεια μιλώ και για τις μικρομεσαίες κυρίως βέβαια εκμεταλλεύσεις και κυρίως ε, για μειονεκτούς περιοχές όπως είναι οι ορεινές περιοχές. Θέλω να πω πάντως ότι εν λόγω έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω γιατί έχει λάβει υπόψη μεσητής εντάσσεται στο πλαίσιο της γνωμοδότησης που ψηφίσαμε στην Επιτροπή των Περιφερειών για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ήταν η ρύθμιση σε σχέση με τις πολύ μεγάλες διακυμάνσεις των προϊόντων, των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Και στην Επιτροπή των Περιφερειών διατυπώσαμε προτάσεις, οι οποίες ελήφθησαν και όλα υπόψη ε, στον κανονισμό Omnibus ε, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, σε σχέση με τη γεωργική πολιτική. Εντάσσεται επίσης αυτή η γνωμοδότηση στις συνολικότερες προτάσεις ε, που είχαν γίνει για την καταπολέμηση του αθέμη του ανταγωνισμού στο πλαίσιο του γεωργοδιατροφικού κλάδου για την ε, ενίσχυση και στο Όμνιμπους ε, και στη γνωμοδότηση αυτή για την ενίσχυση λέγω της δυνατότητας των παραγωγών, των ενώσεων παραγωγών για να μπορούν να προχωρήσουν προς τα εμπρός ως συνομιλητές που θα μπορέσουν να σταθούν απέναντι στον ανταγωνισμό από τι μεγάλε γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Είναι σημαντικό το θέμα, δεν πρέπει να το δούμε απομονωμένο, διότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και σε μια μόνιμη προσέγγιση από πλευρά μα ε, που μα οδήγησε, πιστεύω, σε πρόοδου και είμαι πεπισμένο ότι ανεξαρτήτως των δυσκολιών, διότι η γεωργία δεν είναι μία, υπάρχουν διαφορέ, υπάρχουν διαφορετικά εδάφη. Είναι σημαντικό όμως εμείς οι αιρετοί άρχοντες ε, στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να δείξουμε αποφασιστικότητα για να περασπιστούμε την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι η πρώτη ε, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, σε πλαίσιο ενός σχεδίου ευρωπαϊκού χώρου ταξία. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν οταστικά κέντρα, αλλά ο μιλητής, υπάρχει και σε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκουίντο Μιλάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι θέλουμε δίκαιη, βιώσιμη και κοινωνική γεωργία. Το ερώτημα είναι πώς. Ποια είναι η πορεία για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Εγώ είμαι ένας από τους ε, ε, εισηγητές τόσων ε, τροπολογιών, 115 και σε πολλά σημεία αποκλίνω από τη θέση του εισηγητή, ο οποίο έχει χαράξει μια πορεία για να πετύχουμε του στόχου αυτού, ε, που απέχουν αρκετά από τα πραγματικά συμφέροντα τη ε, γεωργία και τη κτηνοτροφία. Είμαι κατά τη ε, απόλυτη κατάφαση ότι πρέπει να στηρίζουμε την ετήσια παραγωγή μόνο. Επίση, τη απόλυτη μείωση των φυτοφαρμάκων, διότι είναι διαφορετικέ οι σύγχρονε τάσει για την καλή διατροφή ή το πώ προστατεύουμε του καταναλωτέ. Είμαι κατά τη της απόλυτης ε, τοποθέτησης για την ε, κατάργηση των σφαγίων. Όμως θέλω να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε η κοινή αγροτική πολιτική να ξεκινήσει να αλλάζει τις διαδικασίες αυτές, να δημιουργήσει ένα κοινωνικό και οικονομικό ε, μοντέλο το οποίο να επιδιώκει την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών. Ε, δίκαιο δεν είναι μόνο να πληρώνουμε στους γεωργού και κοινοτρόφους την τιμή ε, το τίμημα μάλλον για την ε, περιβαλλοντική ρήπανση, γιατί αυτό αρχίζει να γίνεται παχθέ για τη συγκεκριμένη προβληματική κατηγορία. Και η πολιτική αυτή θα πρέπει να παραμείνει κοινή, αλλά αν θέλουμε να παραμείνει κοινή, δεν χρειάζεται να γίνουμε άκαμπτοι. Άκαμπτοι από την πλευρά τη δίκησης, τη δημόσια δίκησης. Ούτε χρειάζεται να προβλέπουν κανόνε που να είναι υπερβολικά αυστηροί. Χρειάζεται ευελιξία. Είναι βασική συνιστόσα ώστε οι χώρε. Ε, που ε, λαμβάνουν τις αποφάσεις για την κοινή πολιτική ε, να μπορούν να έχουν και κάποια διαλλακτικότητα στη διάθεσή τους, κάποια ευελιξία. Η γνωμοδότηση όπως έχει διαμορφωθεί προς στιγμή δείχνει πολλά σημεία αδιαλαξίας δείγματα διαλαξία. Εδώ λοιπόν στην ψηφοφορία θα φανεί τι θα γίνει με τι τροπολογίε. Θα πρέπει κάποιε να περάσουν για να δούμε τι θα γίνει τελικά με την έγκριση τη έκθεση. Κοιτάζουμε το τι θα γίνει μακροπρόθεσμα. Δεν μα ενδιαφέρει να περάσει η έκθεση αυτή ω προεκλογικό μανιφέστο. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Άρνολτ Χάτσε έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικά σύντομα σημεία. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κρός, τον εισηγητή μας, για την εργόδη προσπάθειά του κατά την εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης. Είναι σημαντικό τη της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πάντως ε, δεν ε, συμφωνώ με αρκετά από τα σημεία της. Για παράδειγμα, δεν ευθυγραμμίζεται με τη θέση της ομάδας μου στο παρελθόν. Επίσης ενθαρρύνει την ε, θέσπιση νέας νομοθεσίας ακόμη πιο έντονη στην ΚΑΠ υπέρ της εξυγχρονισμού, της ψηφιοποίησης, της οικονομίας και ούτω καθεξής. Είναι υπέρ της αύξησης δηλαδή της νομοθετικής ε, ε, ρύθμισης. Επίσης, σε ό,τι αφορά 70.000 ευρώ που είναι το όριο την υποστήριξη των νεαρών αγροτών. Και αυτό αντιβαίνει στο πνεύμα της έκθεσης για τους νεαρούς αγρότες που είχαμε εγκρίνει πριν από δύο χρόνια και που ήθελε να ενθαρρύνει ε, την διείσδυση των νέων αγροτών ε, στη γεωργική δραστηριότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί παραγωγή τροφίμων ε, στην Ευρώπη και γενικώ στον κόσμο. Και μάλιστα έχουμε πρόβλημα και με την εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων. Αυτό είναι παράδεκτο κατά τη γνώμη της ομάδας του ECR. Και η φιλόδοξη αυτή στόχη κατά τη γνώμη της Βρετανικής Αντιπροσωπείας παρά είναι φιλόδοξη σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών από τη γεωργία, τη βιολογική γεωργία, την περιορισμό των φυτοφαρμάκων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και η σύστασή μας είναι ψηφοφορία κατά το δοκούν, κατά συνείδηση, ελεύθερα. Γιατί υπάρχουν πολλά σημεία της ε, γνωμοδότησης που δεν μας βρίσκουν σύμφωνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ραφαέλε Κατάνε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ υπέβαλα ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών για την έκθεση αυτή και προσπέγραψα και άλλε πάρα πολλέ. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλά σημεία τη εκθέση αυτή που δεν με πείθουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει κατά πολύ το περιεχόμενο τη έκθεση με την προφορία στην Ολομέλεια και κυρίω ω προ δύο πτυχέ. Είμαστε Επιτροπή των Περιφερειών. Εκπροσωπούμε ενώπιον των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων τι περιφέρειε και τι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση, τι επαρχίε τη Ευρώπη. Οι γεωργοί που θέλουμε να προασπιστούμε είναι γεωργοί ε, που δουλεύουν στη γη, ε, επιτόπου είναι γεωργία παραδοσιακή, ε, ιστορική των ε, διαφορεών και της ε, ποικιλομορφίας. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε γεωργία ομοιόμορφη βάσει ενό αφαιρημένου ευρωπαϊκού προτύπου. Αυτή είναι η ουσία των περισσότερων τροπολογιών που έχουμε υποβάλει και επαναλαμβάνω, οι περιφέρειες και οι επαρχίες είναι οι βασικοί μας αρμοδιότητες. Και επίσης πρέπει να πω ότι εδώ και λίγους μήνες είμαι υπουργό περιβάλλοντος για την περιφέρειά μου. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό φυσικά αλλά πρέπει τη σχέση μεταξύ γεωργία και περιβάλλοντο να την αντιμετωπίσουμε με τρόπο πολύ ρεαλιστικό, πραγματιστικό. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μια αφηρημένη θεώρηση του τι συμβαίνει ε, στο περιβάλλον και δεν, να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ιδίω για τον τομέα τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Διότι τα αποτελέσματα που θα πετύχουμε θα είναι τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα. Και εδώ η γνωμοδότηση του συναδέλφου ε, Κλάουσκε, και τον ευχαριστώ για τη δουλειά του, έχει, κρόσ, συγγνώμη, ε, έχει σε κάποια σημεία προβάλλει μια σχέση λίγο εξεντερικευμένη για το περιβάλλον και τη γεωργία. Δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα. Επ' αυτού λοιπόν νομίζω ότι στην ψηφοφορία θα πρέπει να αλλάξουμε κατά πολύ πολλά σημεία τη έκθεση για να μπορέσει να περάσει στην τελική ψηφοφορία και να εγκριθεί. Σας ευχαριστώ. Δύο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να πούμε κάτι και για τις κλιματικές αλλαγές και για τη βιοπικιλότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων, καλή διαβίωση των ζώων. Γιατί πλησιάζουμε στο 2020 και θα ήταν λάθος μήνυμα να μειώσουμε, να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας. Γιατί και η Γεωργία εξαρτάται από το κλίμα και τη βιοπικιλότητα. Και οι υψηλέ προδιαγραφέ και τα πρότυπα που απαιτούμε δεν είναι ει βάρο των γεωργών, αλλά προ όφελό του. Γιατί η γεωργία θα επηρεαστεί κατά κύριο λόγο από αρνητικέ κλιματικέ αλλαγέ. Ακριβώ η γεωργία και η κτηνοτροφία θα επηρεαστούν. Οπότε ε, η συρρήκνωση των φιλοδοξιών θα δώσει πολύ λάθο μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο κανεί το λόγο. Οπότε να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την έκθεση του πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία περιλαμβάνει. Ε, Σε ό,τι αφορά ε, τη γεωργία, το περιβάλλον, υπάρχουν όμως ε, κάποια σημεία ε, στην ε, γνωμοδότηση που δημιουργούν κάποια ζητήματα. Ε, σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Πρέπει να πω ότι έχει εδώ και καιρό μεγάλη φορολογική επιβάρυνση και άλλες επιβαρύνσεις ε, και αυτά πρέπει να τα ελαφρύνουμε, όχι να τα επιδεινώσουμε ακόμη περισσότερο. Έχω και συγκεκριμένες τροπολογίες ε, με τις οποίες προτείνω την ελάφρυνση τη φορολογική. Και ανάλογα με το πώς θα ψηφίσουμε σε σχέση με τις τροπολογίες αυτές θα, θα σας δώσω και την τελική μου υπόδειξη για το πώς θα ψηφίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, να, να δούμε τι έχουν να πούν ε, οι συντάκτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι να σας πω. Οφείλω να ομολογήσω ότι με σόκαραν κάποιες παρατηρήσεις που άκουσα. Όταν μου ε, επιπλήττουν γιατί η έκθεσή μου είναι άκαμπτη, ανελαστική και περιλαμβάνει πολλά στραβά σημεία και μερικές φορές υπονομεύω τα συμφέροντα της Γεωργίας, τι να πω. Δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ σουρεαλιστικά αυτά τα σχόλια. Και όταν μου λέτε ότι μερικοί είναι κατά τη αύξηση των ενισχύσεων προς του μικρούς γεωργούς. Θεωρείτε ότι θα διαφωνήσουν οι μικροκαλλιεργητές με την αύξηση των ενισχύσεων προς αυτούς. Επίσης, όταν ζητούμε πιο φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα, θεωρείτε ότι αυτά είναι ανεδαφικά, ουτοπικά. Όταν ήδη βλέπουμε ε, ότι υπάρχουν κλιματικές αλλαγές δεν πρόκειται να δούμε τις αρνητικές συνέπειες σε 10-20 χρόνια. Ήδη τις διαπιστώνουμε. Και πραγματικά για όλα αυτά έχω συγκλονιστεί. Γιατί ως εκπρόσωπος περιφέρειας και ως ερετός περιφέρειας ακριβώς έχω μία άποψη για την πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα. Και αν δούμε τι συμβαίνει στη Γεωργία, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, θα διαπιστώσουμε ότι χρειαζόμαστε κοινού κανόνε, πανευρωπαϊκού. Και όταν λέμε ότι κάποια κονδύλια θα πρέπει να αφιερωθούν για την πράσπιση της βιοπικιλότητας ή για την αναδιανομή Μα λένε ότι είμαστε θεωροβάμενε. Με αυτό προβλέπει ότι κάπου το 80% των ενισχύσεων τη ΚΑΠ πηγαίνουν σε 20% των γεωργών. Αυτό δεν σα σοκάρει. Παρακαλώ, προσέξτε το. Ήδη υπάρχει φοβερή συγκέντρωση των ενισχύσεων. Εμεί το αντίθετο, επιδιώξαμε να συντάξουμε μια ισορροπημένη γνωμοδότηση που θα ανταποκρίνεται στι κλιματικέ αλλαγέ, θα ανταποκρίνεται στι προκλήσει τη κοινωνία και θα έχει μια γνήσια ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό ήταν το ζητούμενο, γιατί αν δεν δώσουμε ευρωπαϊκή διάσταση στην κοινή γεωρική πολιτική, δεν θα έχουμε πια κοινή γεωρική πολιτική, θα πεθάνει η ΚΑΠ. Και το 2027 δεν θα έχουμε πια κοινή γεωρική πολιτική. Αλλά κάποια επενδυτικά μέτρα αριστερά και δεξιά, κάποια περιορισμένη εμβέλεια μέτρα για τι κλιματικέ αλλαγέ. Μέχρι το 2027 όμω θα έχουμε ήδη ε, γίνει μάρτυρη μιας υπερθέρμανσης του πλανήτη και αύξηση θερμοκρασία κατά ένα ή δύο βαθμούς. Το διακύβευμα λοιπόν είναι κοινωνικό. Και επίσης αφουγκραστείτε το συμπολίτη σα τους ε, Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν μια γεωργία εγκύτητας, θέλουν ποιοτικά τρόφιμα, ασφαλή τρόφιμα. Και όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Εμείς τα αναδεικνύουμε. Εμείς τα προβάλλουμε για να καταφέρει ο Γιώργος να βιοποριστεί από το επάγγελμά του, έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Ξέρετε πόσοι γεωργοί ε, αυτοκτονούν. Κάθε τρεις μέρες έχουμε μία αυτοκτονία γεωργού. Επίσης, έχουμε πολλές ε, ασθένειες λόγω της χρήσης κάποιων προϊόντων που πλήττουν κυρίως τους γεωργούς που τα χρησιμοποιούν, τα φυτοφάρμακα. Ε, ζητώ συγγνώμη που φαίνεται ότι χάνω την ψυχραιμία μου. Αλλά ε, με, κατηγόρησαν για δογματισμό. Εγώ αντίθετο πιστεύω ότι η ιδέα ή το δόγμα ότι θα πρέπει να προσπίσουμε κάποια συμφέροντα, αυτό το δόγμα θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη ανακατανομή προκειμένου να δράσουμε προς το συμφέρον των γεωργών και της ανάπτυξης πέθρου και υπέρ του πλανήτη. Ωραία, ολοκληρώσαμε την ε, γενική συζήτηση επί της γνωμοδότησης του κυρίου Κρός και θα περάσουμε στην εξέταση των 304 τροπολογιών. Τις τροπολογίες ενός 4 ψηφίζουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 5 του εισηγητού. Κατά, ε, ποιος είναι υπέρ? Διαγράφει το 5. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ? κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7 του εισηγητού που καταπίπτει το 7α νέο. Ποιος είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 11 του εισηγητού που 11-14 τα διαγράφει. Ποιος είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 15 του εισηγητού που ε, ακυρώνει 15-18. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 του εισηγητού που διαγράφει τα 19 21. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 και 23 που είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ, κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 24. Έχει καταπέσει. 25 το εισήγητο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται 29 υπέρ ή μάλλον όχι, έχει ήδη εγκριθεί Ποιο είναι υπέρ της τροπολογίας 29 κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά vote Τέλος, η ψηφοφορία εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 31 που είναι πανομοιότυπη. με 30 καταπίπτει και αυτή. Τροπολογίε 32 και 33 που είναι ταυτόσιμε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται μάλλον. Τροπολογία 34 του εισηγητού που αντικαθιστά τα 34-36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ κατά εγκρίνεται 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εγκρίνεται 41 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία Le vote est clôturé. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 41. 42 τώρα. Κατά. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πανομοιότυπη ότι είναι με τη 44 οπότε ή 44 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Πάμε στη 45 του εισηγητού που αντικαθιστά τη 45-47. Ποιο είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, 49 και 50 που είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τροπολογία 51, 52 και 53 που επίσης είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικό έλεγχο Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clôturé et la... Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Amendement 51. 51-54. Τις ψηφίσαμε. Μου λένε 54, 55, 56 και 57 είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνονται. 58. Donc, 5, le 58 est devenu Το 58 καταπίπτει. Πάμε στο 59. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 62 έχει αποσυρθεί. 63. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 64 το εισήγητο. Που αντικαθιστά τις 64 ως 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 του εισηγητού. Που ακυρώνει τις 66 ως 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται 72 ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 73 του εισηγητού που ακυρώνει τις 73 και 74 ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 75 ποιος είναι υπέρ Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clôturé. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η τροπολογία. 75. 76 τώρα, που αντικαθιστά την 77 α, υπέρ, μάλλον που ακυρώνει την 77, κατά, απορρίπτεται. 77, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 80 που αντικαθιστά 81-85 υπέρ κατά εγκρίνεται 86 υπέρ κατά απορρίπτεται 87 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Le vote est clôturé. Πέρας, εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 89 κατά εποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία Le Πέρας, η τροπολογία απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά από ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le volet clôturé et l'amendement... Απορρίπτεται. 91. Ταυτόσιμη με την 92. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 94. Ταυτόσιμο με την 95 και την 96. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 97. Υπέρ. Ταυτόσιμο με την 98. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 99. Εάν εγκριθεί η 100 και καταπίπτει, υπέρ, κατά εγκρίνεται 100 Α, ε, 100 και 102 κατά και 101 ταυτόσιμες οπότε φτάνουμε στην 103 υπέρ κατά εγκρίνεται 104 του εισηγητού καταπίπτουν 105 και 106 να υπέρ κατά εγκρίνεται 106 υπέρ κατά εγκρίνεται 107 ταυτόσιμο με την 108 υπέρ κατά εγκρίνεται 109. Καταπίπτει 110. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ισοφορία. Le vote est Πέρας. Εγκρίνεται. 111. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 113. Κατά πίπτουν 114 και 115 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 116 του εισηγητού ακυρώνει την αρχική 116 υπέρ κατά εγκρίνεται 117 α ναι 118 του σιγητού, Κατά τον 119 και 118 αρχική υπέρ. Κατά αγκρίνεται 120 του εισηγητού. Κατά των 121 και 2 υπέρ. Κατά αγκρίνεται 122 κατά εγκρίνεται. 123 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 125 του συγκεκριμένου καταπίπτουν 125 έως 127 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 128. Ταυτόσουμε την 129 και 130 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 131. με τον 132 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le vote est clôturé et... Εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 135. Ταυτόσιμο με την 136. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 137. Ταυτόσιμη με την 138. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 139. Ταυτόσιμη με την 140 και 141. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 142. Καταπίπτουν η 142 του εισηγητή, την αρχική 142 έως 144 υπέρ κατά ηλεκτρονική. Le vote est clôturé et l'amendement est... απορρίπτεται. 142 αρχικό. Ε, με 343 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Clôturé et adopté. Εγκρίνεται. 144. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 145. ίδια με την 146. Και καταπίπτει 147. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 148. 150 καταπίπτει και είναι και ταυτόσιμη με την 149. Ε, Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le Πέρας. Απορρίπτεται. Εκατόν πενήντα. Υπέρ. Κατά. Α, πενήντα ενα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 151. Α, με συγχωρείτε. 152 πήγαμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 153. Οπότε καταπίπτει η 154 ή 155. Υπέρ. Απορρίπτεται. 154 να ψηφίσουμε τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 155. Υπέρ. Α, ταυτόσημη. Ωραία. Ψηφίστηκε. Άρα. 156. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 157. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται.

κατά εγκρίνεται 162 α αποσύρθηκε 162 και καταπίπτει 163 και 164 υπέρ κατά εγκρίνεται 165 υπέρ κατά απορρίπτεται 166 υπέρ κατά απορρίπτεται 167 υπέρ κατά απορρίπτεται 168 υπέρ κατά εγκρίνεται. Κατέπεσε 169. 170 υπέρ. Απορρίπτεται. 171. Κατά. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le vote Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 175. Αποσύρθηκε. 176. Ο εισηγητής, ο εισηγητής προτιμά την 178 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην 179 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 181 της ηγητή υπέρ. Μάλλον αν εγκριθεί από 181 183 καταργού, καταπίπτουν θέλει το λόγο αυτό ο συζητητή, α, όχι αυτό ο συζητητή, αλλά από αυτή την τροπολογία. Ε, αυτή η τροπολογία λοιπόν αφορά του στόχου μείωση των αερίων θερμοκηπίου και στόχος είναι να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη εκδοχή είχαμε ως στόχο του 50%. Εδώ λαμβάνω υπόψη ε, το τι μου είπαν ορισμένοι συνάδελφοι, οπότε ο στόχος πλέον είναι 30%, κάτι που συνάδει, μείωση εννοώ έτσι, των φερμακηπιακών αερίων, κάτι που συνάδει με τους προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των ε, Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία 181 του εισηγητή ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην 184. Όχι, 185 ΠΕΡ. Μάλλον είναι και οι δυο ταυτοσιμε ταυτόσιμες, 84-85. Καρκατά αποχέ εγκρίνονται. 186. του εισηγητή αντί των 186 188 ο εισηγητής θέλει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ θέλουμε την επιφάνεια βιολογικής καλλιέργειας να ορίσουμε. στόχος είναι ανάλογος ε, με αυτό που είπα πριν. Ε, είχαμε βάλει στην αρχή τριπλασιασμό, αλλά άκουσα τους συναντέλφους και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό, οπότε προτείνω διπλασιασμό πλέον. Αλλά πραγματικά να το λάβουμε υπόψη αυτό ότι είναι ένα θέμα δημόσια υγεία, ε, το θέλουν οι καταναλωτέ. Και πραγματικά πρόκειται για σημαντική προσθέμενη αξία για του αγρότε όσοι έχουν προχωρήσει σε αυτό ε, νιώθουν πραγματικά πολύ καλύτερα και το βλέπουν και οικονομικά. Ωραία. Ψηφίζουμε το 186 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. parler aussi. Si c'est Le Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Πηγαίνουμε λοιπόν ε, στην 189 του εισηγητού αντί ε, των 181 192 Συγητή, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Έτυχε τώρα ε, που παίρνω το λόγο τρεις φορές συνεχόμενα. Ίδιο πνεύμα εδώ, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και πάλι αρχικά είχα βάλει 50% μάλλον ήταν υπερβολικό ίσως σε πρώτο χρόνο, οπότε πλέον υποχωρούμε στο 30% είναι στόχος δημόσιας υγείας. Μπορούμε λοιπόν να ε, κάνουμε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μιλάω για πλήρη κατάργηση, αλλά για μείωση 30%. Ωραία, λέω ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε. Oh, στην 193 που είναι ταυτόσιμη την 194 υπέρ κατά απορρίπτονται. Υπάρχει τώρα η 195 του εισηγητού αντί της 195 που καταπίπτει. Αλλά τι υπάρχει εδώ, μια προφορική συμβαστική πρόταση. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητά γι' αυτό. Το κείμενο το έχετε στην οθόνη σας. Ναι, πράγματι, μετά από τις συζητήσεις ε, ε, που είχαμε με τον κύριο Μιλάνα, καταλήξαμε σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, την καλή μεταχείριση των ζώων. Δεν μιλάμε για χορτοφάι και τα λοιπά, μιλάμε για την καλή μεταχείριση των ζώων. Προοδευτικά και συντεταγμένα θέλουμε να προχωρήσουμε στο τέλος, τέλος πάντων, στη μείωση της χρήσης των κλοβών εκτροφής. Άκουσα τους καταναλωτές, άκουσα τους ε, πολίτες της Ένωσης να ζητούν ε, να δοθεί τέλος ε, στην βιομηχανική εκτροφή μέχρι το 2025. Εδώ κάνουμε μια πιο προοδευτική πρόταση, πιο σταδιακή. Σταδιακή πάυση λοιπόν της εκτροφής. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας αυτής, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και έχουμε την 196 και την 197 και την 198 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Και φτάνουμε στην 199 ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Έχουμε τώρα τη 200 του εισηγητή που αφορά στο πρωί 200-203. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και κατά καταπίπτουν οι προαναφερθησει 204 204-205 ταυτόσμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 206 του εισηγητού αφορά τις 206-208 υπέρ. Κατά Εγκρίνεται κατά πίπτων οι προαναφερθήσεις. 210. Ε, πίπτη. Α, με συγχωρείτε. Πήδηξα μια σελίδα. 209 της ηγητού. Αντί τις 209 και 210. Ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 211. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Le vote est clôturé. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία. Και προχωρούμε στην 212 του εισηγητού αντί των τροπολογιών 212 έως 214. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 215 ταυτόσημη με τη 216. Ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 217 και 218 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 219, 220-221 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 222 και 223 ταυτόσιμες ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 224 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 225 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 226 και 27 είναι ταυτόσμες υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Προτείνω να ψηφίσουμε ομαδών της 228 έως και 236 ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνονται. ...237 ψήφι πέρ Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 238. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία. 239. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 240 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 241 που ακυρώνει τη 242. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο vote Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 242. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 243 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 244 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία. 245. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. 246 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 247 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 250 που είναι πανομοιότυπη με τις 251 και 252. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 253 που είναι επανομοιότυπη με την 254. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 256 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 256 ήταν πανομοιότυπη με προηγούμενη, οπότε δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Είμαστε στη 258 τροπολογία, που όμω είναι ταυτόσιμη με τη 259, τη 260 και τη 261. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη 262 υπέρ κατά εγκρίνεται 263 υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 2.64. Ποιος είναι υπέρ. Contre. Adopté. L'amendement. Εγκρίνεται. 2.65 του εισηγητού που καλύπτει την 2.65 και 2.66 τις αρχικές και τις ανεκαθιστά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται 267 υπέρ κατά απορρίπτεται 268 υπέρ κατά εγκρίνεται 269 καταπίπτει 270 qui est Pour. Qui est contre. Adopté. Κατά. Εγκρίνεται. 271 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. Amendement 273. 273 του εισηγητού που αντικαθιστάται 273-1, 275 και ο εισηγητής μας ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια τροπολογία που αφορά τις εκούσιες ενισχύσεις για μείωση παραγωγή σε περίπτωση, της παραγωγής σε περίπτωση κρίσης. Ε, θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο να επεμβαίνουμε εκουσίως, εθελοντικά στην αρχή της κρίσης παρά να αφήσουμε την αγορά να δράσει μόνη της. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, αλλά στην περίπτωση γαλακτοκομικής κρίση το μέτρο αυτό ήταν αποτελεσματικό, παρόλο που εφαρμόστηκε κάπως καθυστερημένα. Πάντως, αν ε, προσπαθούμε καθυστερημένα να διαχειριστούμε την κρίση, δηλαδή να επιφέρουμε λύσεις αφού έχει ξεσπάσει η κρίση, θα είναι πολύ πιο δαπανηρή η διαχείριση. Και νομίζω μια τέτοια πρόταση για την εθελούσια μείωση της παραγωγής ε, συνάντηκε με την έκθεση του Ιουλίου 2008 και με την έκθεση Blanc, ε, για, τη μεγάλη διακύμαση των τιμών. Καλώς. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας του εισηγητού. 273 του εισηγητού.

Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. απορρίπτεται. Αρχική 273 που είναι πανομοιότυπη με την 274. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. 275. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 276. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. L'amendement... Τέλος ψηφοφορίας. 276 ε, τώρα. Ποιος είναι υπέρ. 277, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 278 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le volet clôturé et l'amendement. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία. 280 του εισηγητού που ακυρώνει την αρχική 280. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 281 αποσύρεται. Οπότε ψηφίζουμε από κοινού για τη 282 έως 285. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 286. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Le vote Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 287. 287. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 289 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Le vote est clôturé. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 290. Ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 291 του εισηγητού που ακυρώνει τη 291 την αρχική Ποιο είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 292 του εισηγητού που ακυρώνει τη 292 και 293 υπέρ κατά εγκρίνεται 294. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 296 του εισηγητού που ακυρώνει τη 296 και 297 τις αρχικές. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. 298. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 299 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Le vote est clôturé et... Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 299. 300. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτε ψηφοφορία. La parole, Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Τέλος, εγκρίνεται. L'amendement 301 du rapport. 301 του εισηγητού που αντικαθιστά την αρχική 300. Ο λόγος των εισηγητή. Ευχαριστώ. Είναι η τελευταία τροπολογία μου που αφορά τις ασφάλειες. Αρκετά ευαίσθητο θέμα, αλλά πρότασή μας είναι να πούμε ότι προτιμούμε να ρυθμίσουμε τις αγορές παρά να περάσουμε από τις ασφάλειες. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρόκειται για ένα σύστημα που εφαρμόστηκε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και από τα 5 δισεκατομμύρια που στήχησε στο δημόσιο κοροβανά, μόνο 0,2 δισεκατομμύρια επέστρεψαν στους γεωργούς. Όλα τα υπόλοιπα πήγαν στους ασφαλιστές. Οπότε, ναι, στις ασφάλειες για τις κλιματικές, υγειονομικές, ε, ε, ατυχίες, αλλά για τα θέματα της, των αγορών καλύτερα να ρυθμίζουμε τις αγορές παρά να παραπέμπουμε το θέμα της ασφάλειας. Και κάτι τέτοιο ευθυγραμμίζεται και με προηγούμενη μας έκθεση. Καλώς ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 300 του εισηγητού. Κατά. Εγκρίνεται. 302. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται 303 που αντικαθιστά 304 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται οπότε ψηφίζουμε την 304 υπέρ κατά εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ποιος είναι υπέρ της γνωμοδότησης Α, κάποιοι ζήτησαν το λόγο. Δύο λεπτά, ευχαριστώ. Δεν, Δεν μου χρειάζονται δύο λεπτά. Λίγα δευτερόλεπτα μόνο. Να πω ότι η Ιταλική αντιπροσωπεία σκέφτηκε, θεωρεί ότι κάποιες τροπολογίες που εγκρίθησαν από τον εισηγητή, από τους συντάκτη γνωμοδότησης και υπερψηφίστηκαν μεν αλλά άλλα θέματα δεν έγιναν δεκτά και γι' αυτό η τελική Αντιπροσωπεία θα κρατήσει τάση αποχής στην τελική ψηφοφορία. Μάλιστα. Άλλος κανείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν την τελική ψηφοφορία θα ήθελα να σας ζητήσω να ελέγξετε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της ε, τροπολογίας 54, 56 και 57 που ήταν πολύ σημαντικές τροπολογίες γιατί μιλούμε για την ε, εξίσωση των ε, στρεματικών ενισχύσεων και κρίνω σωστό να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτές τις τρεις τροπολογίες. Τελείωσε η ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε μεμονωμένες τροπολογίες. Ένας ακόμη συνάδελφος ζήτησε το λόγο κύριος Άτζο Παρ. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να συστήσω να υπερψηφίσουμε τη γνωμοδότηση μετά τις ψηφοφορίες για τις τροπολογίες. Μάλιστα, άλλος κανείς. Οπότε, τελική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της γνωμοδότησης του κύριου Κρός, όπως έχει τροποποιηθεί. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και μπράβο σας ε, κύριε Κρός. Συγχαρητήρια και σε εσά και στο επιτελείο σας. Και τώρα παρακαλώ τον πρώτο μας αντιπρόεδρο να πάρει τη σκητάλη. Ελπίζοντας ότι στις επόμενες ψηφοφορίες οι τροπολογίες θα είναι πολύ λιγότερες.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 Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so he is not there. Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies. and Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. If a few of you need to have a short break. Αν χρειάζεστε όμως ένα σύντομο διάλειμμα, Μπορείτε να αποχωρήσετε για λίγο. Έχουμε ακόμα αρκετέ γνωμοδοτήσει, αλλά δεν είναι πολύπλοκε και δεν έχουμε και τόσε τροπολογίε. Επόμενη έκθεση, ε, γνωμοδότη καλύτερα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ο Σίμω Πούτ Ιφερέρ, ο εισηγητή. Θα ακούσουμε την ε, παρουσίαση αλλά θα παρακαλέσω τους εισηγητές να είναι σύντομοι από εδώ και πέρα στις ε, εισαγωγικέ παρατηρήσεις για να ολοκληρώσουμε γρήγορα και να διεκπαιρεώσουμε τα θέματα της διάταξης εγκαίρως. Ήσυχα. Παρακαλώ ησυχία και συνεχίζουμε. Δίνω το λόγο στον εισηγητή μας. Θα μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Κύριε εισηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο πρόεδρος ε, της ε, περιφερειακής κυβέρνησης Βαλένθια δεν μπορούσε να είναι εδώ. Ε, θα το ήθελε παρόλα αυτά, τον αντικαθιστώ εγώ. θα να σας πω ότι εδώ και καιρό αυτό το ταμείο όταν πρώτο εμφανίστηκαν τα προβλήματα και οι ανάγκες προσαρμογής της παγκοσμιοποίηση για κλάδους και για περιφέρειες που ήταν στην πρώτη γραμμή ε, αυτής της παγκοσμιοποίησης. Ο στόχος ήταν να αντιμετωπιστούν ε, οι κρίσιμες αυτές καταστάσεις, ιδίως για τους εργαζομένους ε, στους κλάδους, ε, στις περιοχές αυτές, για να τους προστατεύσουμε τους εργαζομένους από τις απειλές και ιδίως πλέον ευάλωτους. Πρέπει να σας πω ότι εμείς καταγόμαστε από μια περιοχή περιοχή η οποία χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποίησε πάρα πολύ, αξιοποίησε πολύ αυτό το ταμείο. Επομένω, γνωρίζουμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται και θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένα αποτελεσματικό και αναγκαίο εργαλείο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε απορρόφησή του από άλλα ταμεία ή από οποιαδήποτε με οποιαδήποτε κατάργησή του. Θέλω να σας πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά με θετικά βήματα, υπό ποια έννοια. Ε, συμφωνούμε ότι πρέπει όλο και περισσότερο να βαδίσουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης των ε, προβλημάτων, να τα προκαταλαμβάνουμε και να προκαταλαμβάνουμε καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν σε διάφορους ε, κλάδους και σε διάφορες περιοχές. Επίσης, όπως σας έλεγα, υπάρχουν διαφορετικές πραγματικότητες ανάλογα με την περιφέρεια, ανάλογα με τον οικονομικό κλάδο. Αυτό που εμείς λοιπόν κυρίως υποστηρίζουμε είναι η μεγαλύτερη ευελιξία για να ληφθούν υπόψη αυτές οι διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις ό,τι αφορά τους μηχανισμούς, τα εργαλεία, το χρόνο και τον αριθμό των θυγωμένων σε κάθε περίπτωση. Και η ευελιξία αυτή είναι αναγκαία για έναν ακόμη λόγο. Αν δηλαδή αρχικά, γιατί εγώ ήμουν στο Κοινοβούλιο όταν ε, πρώτο ξεκίνησε να συζητείτε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Αν είχαμε εστιάσει τι συζητήσει μα τότε σε επιπτώσει τη παγκοσμιοποίηση, άνοιγμα του διεθνού εμπορίου, πώ επηρεάζονται οι διάφοροι κλάδοι, αυτέ ε, οι καταστάσει σήμερα έχουν να κάνουν και με την ε, κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση, την νοημοσύνη και με πολλούς άλλους παράγοντες που καθιστούν απολύτως αναγκαία την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού που επίσης πρέπει να είναι και ευέλικτος κατά την άποψή μας για να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Κάλαμπουικ στη θέση του κυρίου Πούτς. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις. Περνούμε λοιπόν ευθύ αμέσω στην εξέταση των τροπολογιών. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Είναι approved. Οι περισσότεροι είναι υπέρ, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Against. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά A few majorities Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Thank you against. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Αν εγκριθεί κατά πίπτη 8 ψήφι υπέρ της 7. Ουδής. Κατά. Είναι κατά ψηφία λοιπόν. Απορρίπτεται. Πάμε στην 8 υπέρ. Κατά. Ουδής εγκρίνεται. Τροπολογία 9 ψήφι υπέρ. Against. Κατά. Ουδής εγκρίνεται. Τροπολογία 10 ψήφι υπέρ κατά κατά οι περισσότεροι απορρίπτεται τροπολογία 11 ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 12 ψήφι υπέρ κατά απορρίφθηκε τροπολογία 13 υπέρ λίγη Κατά. Πολύ. Άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Η περισσότερη κατά, άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Η περισσότερη κατά απορρίπτεται. 16. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Κανένας κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, λίγη. Η πλειοψία είναι υπέρ, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 19, ψήφι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 20, ψήφι υπέρ, κατά, Ουδής εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Όπως τροποποιήθηκε ψήφι υπέρ της γνωμοδότησης κατά ένας. Άρα η πλειοψηφία είναι υπέρ, εγκρίνεται συγχαρητήρια. Και έχετε το λόγο κιόλας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Απλά να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη. Να ευχαριστήσω και τις οργανώσεις και άλλους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Να ευχαριστήσω φυσικά και τους εμπειρογνώμονες που μας βοήθησαν στην εκπόνηση της έκθεσης. Ωραία λοιπόν. Και ευχαριστούμε και εσάς και τον αρχικό εισηγητή, τον καθηγητή τον κύριο Πούτς. Περνάμε τώρα στην επόμενη γνωμοδότηση είναι η συγγετρία κυρία Φόρτ από το ΚΟΡΚ, μέλος του Κομιτιακού Συμβουλίου. Παρακαλούμε, ελάτε κι εσείς εδώ με τον εμπειρογνωμονά σας, στο Προεδρείο μας. And it's about the single market program. Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Έχουμε περίπου 20 τροπολογίες να κοιτάξουμε μαζί. Γεια ελάτε. Okay, Madam Ωραία. Κυρία εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη Ευρώπη. Έχει φέρει τεράστια ωφέλη στου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι επιχειρήσει και εταιρείε. Έχει δημιουργήσει χιλιάδε θέσει εργασία για μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών, ενδυνάμωσή του, για ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κυρίω των μικρομεσαίων και έχει επιτρέψει στον κόσμο να ζει και να εργάζεται, να, να φυτά εκεί που επιθυμεί. Με την πραγματική ε, υλοποίηση πραγματικών ε, προτύπων και τα στην ψηφιακή εποχή. Με τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ επίση και τη συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την σωστή διαμόρφωση αποφάσεων σε πολλού πολιτικού τομεί. Αυτά είναι στην καρδιά τη ε, οικονομική ε, και πολιτική ολοκλήρωση τη Ευρώπη που αφορά πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε και 4 εκατομμύρια εταιρείε. Χάρη στην ενιαία αγορά, ο κόσμο, τα αγαθά, τα εμπορεύματα και το χρήμα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ευρώπη, σχεδόν το ίδιο ελεύθερα σαν να επρόκειτο για την ίδια χώρα. Και ε, εκατοντάδε τεχνικοί κοινωνική, γραφειοκρατική και διοικητική φραγμή στην ελεύθερη κυκλοφορία και το ελεύθερο εμπόριο έχουν αρθεί, ώστε οι ροέ αυτέ να γίνουν ευκολότερε. Οι ε, εταιρείε μπόρεσαν να αναπτυχθούν ανταγωνιστικά με τη μείωση των τιμών και μεγαλύτερη προσφορά για του καταναλωτέ. Η αγορά θα πρέπει όμω να συνεχίσει να ε, προσαρμόζεται σε ένα μετάβολο περιβάλλον. Με την ψηφιακή επανάσταση, με τι επιπτώσει τη παγκοσμιοποίηση. Αυτή τουλάχιστον είναι η απειλή που επικρέμαται μετά την ε, απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Brexit να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις απρόβλεπτες συνέπειες για την ενιαία αγορά γιατί είναι τεράστια πρόκληση και για την επιβολή και την ε, ε, τήρηση της νομοθεσίας. Το να προβλέπει κανείς κανόνες είναι ένα πράγμα, το να τους τηρεί στην πράξη είναι κάτι διαφορετικό και να λειτουργούν. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς θα στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στην ενιαία αγορά. Το τονίζω αυτό στην εκθεσή μου, τονίζω τη σημασία του ρόλου, τους, του ρόλου τους και το πόσο σημαντικό είναι να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς και στα ωφέλη της ενιαίας αγοράς. Στο σημείο 4 Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, επιτρέψουμε ε, ό,τι βοήθεια παρέχουν τα κράτη-μέλη και μετά το 2021 να την ενισχύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να υπάρχει επίσης ε, ψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για την για το EEN, το πρόγραμμα αυτό, όπου θα πρέπει στην ενιαία αγορά, ιδίως στον χρωματοπιστωτικό τομέα και δεδομένου του αντικτύπου που μπορεί να έχουν οι εσφαλμένε αποφάσει στην καθημερινότητα των πολιτών, θα πρέπει εδώ να λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να είμαστε βέβαιοι ότι οι εταιρείε αυτέ δρούν ανεξάρτητα και ε, στηρίζονται από, την, το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών. Η διακυβέρνηση τη κοινή αγορά είναι επίση ζωτική σημασία και οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ μπορούν να συμμετέχουν. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την ενιαία αγορά έχει ε, ενταχθεί ολιστικά στις τοπικές ε, συνθήκες και προϋποθέσεις. Αυτά τα εξετάσαμε στο επίπεδο των δημόσιων προμηθειών, των εργαλείων ε, διακυβέρνησης και τις προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να φτάσουμε στους πολίτες το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και επίση το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι το καλύτερο επίπεδο για να προσφέρουμε καθοδήγηση στου πολίτε που χρειάζονται καθαρτήρες γραμμές εκεί που ζουν. Ευχαριστώ επίσης πολύ τους συναδέλφους από το ΕΛΚ για τις τροπολογίες τους και θα ήθελα να ολοκληρώσω με αυτό το σχόλιο. 25 χρόνια έχουν περάσει από αυτό που δημιουργήθηκε το πρόγραμμα για την ενέργεια αγορά. Καταφέραμε να ε, εξαλείψουμε πολλούς φραγμούς οι πολίτε έχουν ωφεληθεί. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Όμω πρέπει να συνεχίσουμε για να βελτιωθεί η λειτουργία τη ε, ενιαία αγορά και να συνεχίσουμε να έχουμε απτά ωφέλη για του πολίτε, τι επιχειρήσει μα ε, και ε, τι εταιρείε μα. Θα πρέπει στι μελλοντικέ γενιέ να κληροδοτήσουμε μια ελεύθερα κυκλοφορούσα και εύρωστη ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Συγκετρία. Υπάρχουν ε, παρεμβάσεις. Κανείς. Πολύ ωραία. Περνάμε στις τροπολογίες. Περνάμε με την 1R της εισηγήτρες δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Κανείς αποχές. Δίνεται η 2 καταπίπτει. 2R της εισηγήτριας. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται δύο, οι δύο καταπίπτει λοιπόν, οι δύο αρχικοί. Ε, η τρία υπέρ, κατά. Η πλειοψηφία είναι υπέρ, εγκρίνεται. Καλά, ας ψηφίσουμε και ηλεκτρονικά. Τρία. Okay, we close the vote. Πέρας. 31, 26 κατά. Εγκρίνεται. Η 4 καταπληκτή. Αφού εγκρίθηκε η 3. Ψηφίζουμε μαζί 5, 6, 7. Μπλοκ υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Τροπολογία της εισηγήτριας 8R υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Κανείς εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει 9 υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Εγκρίνεται 10. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά απορρίπτεται 12 της εισηγήτριας υπέρ κατά άρα η πλειοψηφία είναι υπέρ οπότε εγκρίνεται 12 καταπίπτει να ψηφίσουμε μαζί τις 13 έως 17 unblock υπέρ ψηφίστε τώρα παρακαλώ κατά κανείς εγκρίνονται 13, 14, 15, 16, 17 18 υπέρ κατά υπέρ. Α, οι περισσότεροι άρα εγκρίνεται 19 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και μετά τελική ψηφοφορία για ολόκληρη την ε, γνωμοδότηση, όπως τοποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Κανείς. Αποχές. Καμία. Ομόφωνη έγκριση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, κυρία Ντέιντ Φόρντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το χάρηκα πολύ. Φανταστική δουλειά. Μπράβο σας. Οκ. Okay. Μάλιστα. Περνάμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη γνωμοδότηση. και καλώ τον Αντιπρόεδρο Αμπράμοβιτς να προεδρεύσει για να μπορέσω εγώ να λάβω το ρόλο του συντάκτη της Ladies and gentlemen, move on. Περνάμε κυρίε και κύριοι στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για το 2021-2027. Με χαρά μου να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μάρκο Μάρκουλα, για την παρουσίαση της γνωμαδότησής του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ε, τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, τον καθηγητή Τανατούκεν που ήταν ο εμπειρογνώμονάς μου για το θέμα αυτό και γνωρίζει καλά αυτά τα θέματα και στο παρελθόν όταν εργαζόταν στο γραφείο μου η εμπειρογνώμονας επίσης τον Αλεξάνδρ Πόποβατς και στη γραμματεία θερμά ευχαριστώ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μου έδωσαν γιατί ήδη τον Ιούλιο είχαμε την πρώτη συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή του για το θέμα αυτό, οπότε είχαμε στενή συνεργασία ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και σε επίπεδο διευθύνσεων. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικά νευραλγικά σημεία της έκθεσης. Μετά από μία δεκαετία, θα έλεγα, πειραματισμού, η έφης πόλεις ε, με τις ψηφιακές υποδομές περνάνε σε μία νέα φάση. Και παρόλο που είναι ένα τμήμα μόνο του συνολικού πλαισίου, δείχνει ότι η ψηφιοποίηση δίνει στις πόλεις ε, μεγάλες λύσεις και βελτιώσεις. Σίγουρα οι ψηφιακές λύσεις είναι οι πιο ισχυρές και οικονομικά ε, συμφέρουσες λύσεις για την βελτίωση των δραστηριοτήτων των πόλεων. Και ένα παράδειγμα τέτοιε δραστηριότητε που στηρίξαμε και την έκθεσή μα, μάλιστα, και που εφαρμόζεται σε πολλέ καθευθυντήριε γραμμέ τη πολιτική, είναι η ψηφιοποίηση των διασκέψεων κορυφή των πόλων. Αυτό που σα ανέφερε πριν ο κύριο Λάμπερτ και το είπε και στην εισαγωγική του ομιλία κατά την άραξη της Ολομέλειας. 41 πόλεις και κυρίως οι δήμαρχοί τους συμμετείχαν με τους βοηθούς τους στην ε, διάσκεψη κορυφής ε, των ψηφιακών πόλεων που οργανώθηκε από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, από την Γενική Διεύθυνση Growth της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και μάλιστα χθε πολλοί δήμαρχοι συνέχισαν το έργο τους και τις συναντήσεις τους στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης κορυφής. Και πριν περάσω τη μητρική μου γλώσσα τα φιλαδικά θα ήθελα να πω να ευχαριστήσω θερμά φυσικά επαναλαμβάνω του συνεργάτε μου και να πω ότι η ψηφιοποίηση διαδραματίζει κέριο ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων όπως ε, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και στην υλοποίηση και των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να πρωτοστατήσουν παγκοσμίω, να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να αναλάβουν ε, τις ευθύνες τους ε, και στο μέλλον. Και σίγουρα ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, γιατί μόνο σε συνεργασία και με αποφασιστικότητα θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας της ψηφιοποίησης. Κατά την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να έχουμε λειτουργικότητα σε όλη την Ευρώπη και φυσικά ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε εταιρικέ σχέσεις μεταξύ των πόλεων και πολλές εταιρικέ σχέσεις σε τοπικό επίπεδο μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων ε, ή επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων. Χρειάζονται τέτοιες πολυμερείς εταιρικέ σχέσεις ε, μεταξύ των περιφερειών και μεταξύ των πόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη γνωμοδότησή μου επισημαίνω την ανάγκη για ποιοτικά δεδομένα και την συγκέντρωση επαρκών δεδομένων ώστε η τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των ε, πόλων να γίνει πραγματικότητα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του ρόλου των νέων προγραμματιστών γιατί έχουμε δημόσια πρόσβαση όλο και περισσότερο δεδομένων και προωθούμε τέτοιου είδους δημόσια πρόσβαση. Στην γνωμοδότηση αναδεικνύουμε και το ρόλο των ε, περιφερειών, των δήμων και κοινοτήτων και ζητούμε ένα, τη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των ψηφιακών κόμβων που θα έχει πανευρωπαϊκή εμβέλεια, ώστε κάθε περιφέρεια να έχει το δικό της κόμβο ψηφιακής καινοτομίας, κάτι που είναι απαραίτητο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να έχουν έντονα ευρωπαϊκή διάσταση. Μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε την επιθυμητή ανάπτυξη. Έχουμε κάνει πολλές διευκρινήσεις στη γνωμοδότηση λέγοντας ότι θέλουμε τέτοιους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας τέτοιους θύλακες που ε, η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται από πολλούς παράγοντες, πολλούς φορείς σε συνεργασία και με νομική πλαισίωση. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και ομίλους. Επίσης, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα τόσο ισχυρό πακέτο που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση, την έρευνα και την καινοτομία και μάλιστα σε όλα τα σημαντικά και μεγαλεπίβολα ευρωπαϊκά προγράμματα Κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργεί μια ολοκλήρωση. Επίση, η χρηματοδότηση είναι σημαντικό θέμα που συζητάτε στα πλαίσια του ρημαρούς διαλόγου. 9,2 δισεκατομμύρια είναι το αρχικό κονδύλιο. Είναι σημαντικό για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να αναλάβουμε παγκοσμίω τις ευθύνες μας ως ε, βασικός παραγοντας της ψηφιοποίησης. Μία, ψηφιο... μία τροπολογία έχω μόνο, γιατί με καλύπτει κατά άλλα η γνωμοδότηση και νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολη η διεκπαιρέωσή της. Στην τροπολογία επισημαίνω περισσότερο αυτά τα σημεία από ό,τι στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση μετά την εισαγωγή που μας έκανε ο συντάκτης γνωμοδότησης, αν υπάρχει ενδιαφέρον φυσικά. Αν όχι, περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία των τροπολογιών. Αλλά μία τροπολογία έχουμε μόνο από, τον, από το ECR και τον εισηγητή. Από το ECR μάλλον και ο εισηγητή, ο συντάκτης γνωμοδότης έχει καταθέσει και δική του τροπολογία. Ψηφίζουμε την τροπολογία παριθμών 1 του εισηγητού του κ. Μάρκουλα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης μετά την τροποποίηση. Ωραία. Υπέρ, κατά. Κανείς. Αποχές. Ούτε καμία αποχή. Οπότε συγχαρητήρια κύριε Μάρκουλα. Με θερμό χειροκρότημα γιατί ομόφωνα εγκρίνεται η γνωμοδότησή σας και να σας ανακοινώσω τώρα ότι οι δύο τροπολογίες, η καταρχήν του Ματέο Λουίτζι Μπιάνκη για το Ευρωπαϊκό σώμα και την νέα στρατηγική για την όλα αναβάλλεται για αύριο, το ίδιο και η γνωμοδότηση του κυρίου Αντρές Γιάντλα για το διαστημικό πρόγραμμα αναβάλλεται για αύριο, οπότε μια καλή είδηση. Για σήμερα διεκπαιρώσαμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω επίση ότι η Αυστριακή Αντιπροσωπεία θα ήθελα να σας προσκαλέσει την δεξίωση που οργανώνει στο Άτριο της Επιτροπής των Περιφερειών. Όσοι έχουν απομείνει λοιπόν, ε, έχουν, είναι άξιοι, αντάξει αυτής της δεξίωσης της ε, Αυστριακής Προεδρίας. Καλό σας βράδυ.